Κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Οι αποφάσεις των συντονιστών από τη χθεσινή του συνεδρία σας έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι θα εγκρεθούν και προχωρούμε στην ανταλλαγή ε, πληροφοριών, απόψεων μάλλον, για το θέμα των θα, θα ψηφίσουμε μάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών στις ε, διασυνοριακές ε, οδικές μεταφορές με την κυρία Γιάννα Σάντερος Ξεκινάμε δοκιμαστικά πρώτα την ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Ώρα λειτουργούν σωστά από ό,τι βλέπω. να υπάρχουν και ωραίες εκπλήξεις στη ζωή ενίοτε. Και πάμε στην υπαριθμόν 11 τροπολογία υπέρ διανατάσεως παρακαλώ. Κατά. Απερίφθη. 12 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη υπαριθμών 6 υπέρ κατά άποχες απερίφθη 7 υπέρ υπέρ κατά άποχες απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη υπαριθμών 1 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστικά θα γίνει η τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά και ονομαστικά. Αρχίζει. Από τη σωστή γωνιά βλέπω έρχονται πάντα παρατηρήσεις. Ωραία τώρα, διορθώσαμε τον αριθμό των ψηφισάντων. Έχουμε 44 ψήφισαν, 36 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ την εισηγητρία. Και τώρα έχουμε το νομοθετικό ψήφισμα παρακαλώ, ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εψήφισαν 44. 34 υπέρ, 7 κατά, 3 αποχές. Και τώρα πρέπει να κάνουμε μια ψηφοφορία για τη με το Συμβούλιο. Ηλεκτρονικά και πάλι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 35 υπέρ. 7 κατά, μία αποχή. Mm. Η επόμενη ψηφοφορία. Σχέδιο πρότασης για απόρριψη του σχεδίου κανονισμού για την κατάταξη των σοβαρών παραβιάσεων των κανόνων τη Ένωση, οι οποίε ενδέχεται να οδηγούν στην απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστία του οδηγικού μεταφορέα. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτη τροπολογία ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Υπέρ. Ψήφισμα, συγγνώμη. Ψήφισμα, πρώτο ψήφισμα. ΕΛΚ Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Κατά. Αποχές. Καλά, ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέραστη της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 11 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται και ως εκ τούτου καταπίπτουν τα λοιπά ψηφίσματα. Αυτά με τις ψηφοφορίες. Διακόπτουμε τώρα για μερικά λεπτά μέχρι να έρθει η κυρία Μπούλτς.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 Hm?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 Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Βιολέτα Μπούλτς η οποία μας έχει έρθει μαζί με τον κύριο Ματσάρο, Γενικό Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΜΟΥΒ. Καλώς ήρθατε και είναι και η πρώτη φορά. Επίσης θέλω να καλωσορίσω μια ομάδα δημοσιογράφων από την Αυστρία προσκεκλημένων του κυρίου Σμιτ. Σας εύχομαι καλό, το καλώς ήρθατε και ελπίζω να είναι και ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση για σας. Είναι η πρώτη φορά που η κυρία Μπούλτσο ε, έρχεται να μας δει ύστερα από την ανάληψη των καθηκόντων της ως Επιτρόπου. Έχετε το λόγο κυρία Μπούλτσο. Α, σε Ευχαριστώ πάρα πολύ. Morning everyone and best regards from my entire team. Καλημέρα σε όλους. Ήταν ε, πολύ συναρπαστική αυτό το πρωινό και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε με πολύ επικοδομητικό τρόπο όλο το πρωινό. Είμαι πολύ ευτυχής που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια από τις σκέψεις μου και να σχολιάσω και κάποια από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Και ειλικρινά σας λέω χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και ελπίζω πως θα έχουμε πολύ καρποφόρα συνεργασία κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Όπως μάλλον θα θυμάστε, στη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον αυτής της Επιτροπής μόλις πριν από έξι εβδομάδες και έχω την αίσθηση ότι πέρασε ήδη ένας χρόνος, ε, δεσμεύτηκα να συνεργαστώ στενά με καθέναν από εσά και να Είμαι εγώ και η ομάδα μου διαθέσιμη ώστε να έχουμε τακτικές αναφορές και ενημερώσεις για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις δικές μου ε, αρμοδιότητες. Ελπίζω, ε, την τελευταία φορά είχαμε καρποφόρα συνεδρίαση στο Στρασβούργο και ελπίζω πως έτσι θα συνεχιστούν τα πράγματα. Για μένα το πιο σημαντικό κίνητρο για να συναντώμε μαζί σας είναι ότι αναπτύσσεται έτσι η εμπιστοσύνη. Κατανοούμε ότι βρισκόμαστε από την ίδια πλευρά ότι... και ότι θα πρέπει να επενδύσουμε το χρόνο μας στην προετοιμασία των διαφέρων γράφων ε, μαζί έτσι ώστε να οδηγούμεθα σε επιτυχή ολοκλήρωση γιατί είναι κρίμα να σπαταλάμε χρόνο για να και τελικά να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος της προετοιμασίας. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι πολύ ευτυχής που ανταποκρίνομαι στη σημερινή σας πρόσκληση κύριε Κράμερ και να έρθω και πάλι ενώπιόν σας και να ανταλλάξω μαζί σας τις απόψεις μου για το πλάνο επενδύσεων που υιοθέτησε η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα. Ιδιαίτερα τι σημαίνει αυτό το πλάνο το επενδυτικό για τον τομέα των μεταφορών. Να εκφράσω την πλήρη μου υποστήριξη καταρχήν στο πρόγραμμα 315 δις ευρώ που στόχο έχει την προώθηση των θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα είδος ε, δομημένης ε, παρουσίασης ε, των ωφελών για τις μεταφορές θα τονίσω τους τρεις βασικούς πυλώνες που είναι κομμάτι αυτού του επενδυτικού Ταμείου των 315 δις. Πρώτον, δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, δηλαδή χρήμα. Τα, η θέσπιση ενός αξιόπιστου προγράμματος προετοιμασίας προγραμμάτων ε, μαζί με ένα πρόγραμμα ε, αρρωγής. Καταφέραμε, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να φτιάξουμε ένα καλό πρόγραμμα, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς βοήθεια δεν θα έχουμε και καλά projects. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα ίδια τα projects, αλλά και για το ε, εργαλείο αυτό, το μέσο αυτό βοήθειας. Ε, φιλόδοξος οδικός χάρτη είναι ο τρίτο πυλώνα για τη βελτίωση του ρυθμιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Ε, ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα. Οι ιδιώτε επενδυτέ, αν δεν υπάρχει προβλεπόμενο και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν επενδύουν. Ο τρίτος πυλώνας λοιπόν είναι εξίσου σημαντικός. Χρήματα, ε, προγράμματα και ρυθμιστικό περιβάλλον νομοθετικό περιβάλλον και τώρα θα εστιάσω στο τρία αυτά στοιχεία ώστε να υπογραμμίσω τη σημασία τους, την ιδιαίτερη σημασία τους για το τομέα των μεταφορών. Και ελπίζω πως θα είμαι σε θέση να σας ε, μεταδώσω τον δικό μου ενθουσιασμό. Οι επενδυτικέ ανάγκε στι μεταφορέ είναι τεράστιε. Σύμφωνα με μελέτε που έχουν γίνει στους, για του 9 ευρωπαϊκού διαδρόμου, πάνω από 75 δι ευρώ χρειάζονται ετησίω. Μόνο και μόνο μιλάμε για τους διαδρόμους που είναι κομμάτια του δικτύου TEN-T. Δεν έχουμε κάνει τη δουλειά μας ακόμα λοιπόν, ακόμα και αν έχουμε το επενδυτικό πλάνο των 315 δις, που ακούγεται καλούτσικο, αλλά χρειάζονται και περισσότερα. Έπειτα, ε, οι επενδύσει ε, που χρειάζονται είναι εξαιρετικά ψηλές για τις καθαρότερες μορφές ε, μεταφορών, δηλαδή του σιδηρόδρομου και τι εσωτερικέ πλωτέ οδού, εκεί όπου λείπουν κομμάτια ή εκεί που δημιουργείται συμφόρηση πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, ιδιαίτερα στα σύνορα, για να έχουμε πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών. Έπειτα, εγκατάσταση των ε, σημείων ε, ε, φόρτισης για τα ηλεκτρικά, ηλεκτροκινούμενα οχήματα ή η εγκατάσταση LNG, δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικά. Δεύτερον, οι επενδύσεις στην αστική κινητικότητα είναι μαζικές γιατί εκεί υπάρχει περισσότερη κίνηση και οι περισσότερες εκπομπές. Οι υποδομές για τη δημιουργία νέων στόλων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να καταστήσουν τις πόλεις μας ευφιέστερες και πρέπει ήδη να δημιουργηθούν. Τρίτον, θα πρέπει να προσαρμοστεί το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν λοιπόν e e, ευφυή συστήματα μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υφιστάμενες και τις μελλοντικέ υποδομές και να εξυπηρετήσουν πραγματικά τις ανάγκες των χρηστών, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στατικικές Επενδύσεις που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι λοιπόν μεγάλη σημασία για τις μεταφορές καθώς θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ώστε να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες τις οποίες μόλις αναφέρθηκα. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι θα συμπληρώσει και δεν θα αντικαταστήσει τα μέσα που ήδη υπάρχουν, όπως η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το Ταμείο Συνοχής ή τα δάνεια της ΕΤΕΠ, όπου το τομέας των μεταφορών είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους. Με δυνατότητα ανάληψης κινδύνου 21 δις ευρώ, αυτό το νέο μέσο θα στοχεύσει σε πιο επικίνδυνα προγράμματα, πιο επισφαλή προγράμματα από ότι αυτά που έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι τώρα από την ΕΤΕΠ. Επίσης θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ειδών επενδύσεων που δεν έχουν πρόσβαση στις επιδοτήσεις της Ένωσης ή που έχουν περιορισμένη πρόσβαση ε, σε ε, αναλογία προς τις ανάγκες τους. Ας πούμε, ολοκλήρωση ε, οχημάτων με FEE e και καθαρά συστήματα μεταφορών, η e RTMS, η Caesar, τα σημεία γρήγορης ε, φόρτισης, για να αναφέρομαι κάποια. Θα εστιαστεί στα πιο όρημα προγράμματα που μπορούν να ε, ξεκινήσουν εντός των επομένων τριών ετών. Η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, στην οποία συμβάλλατε πολύ για να φτιαχτεί, θα χρησιμοποιήσει το το νέο επενδυτικό ταμείο για να αναπτύξει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα από το νέο ταμείο θα μπορέσουν να καλύψουν ευρύτερου κινδύνου και να ε, κινητοποιήσουν καλύτερη μόχλευση προσελκύοντας πιο πολλέ επενδύσεις με μια αναλογία που αναμένουμε να είναι 1 προς 15 και σε ορισμένε περιπτώσει και ακόμη περισσότερο. Το 10% λοιπόν του προϋπολογισμού του CF που συμβάλλει στην ευρωπαϊκή εγγύηση δεν σημαίνει καμιά αλλαγή όσον αφορά τις προτεραιότητες του ΤΕΝΤΗ και της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη όπως ορίστηκαν αρχικά. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Με έναν ισχυρό προϋπολογισμό στο ΣΕΦ υπάρχουν αρκετές επιδοτήσεις για προγράμματα που διαφορετικά δεν θα χρηματοδοτούνται, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μεγάλα διασυνοριακά προγράμματα και τις συμφορήσεις, ε, τα μποτιλιαρίσματα στους διαδρόμους TNT. Αντιθέτως, τα προγράμματα TNT προτεραιότητας τώρα θα είναι επιλέξιμα και για τις δύο επιδοτήσεις, είτε από το ΣΕΦ και από το χρηματοδοτικό μέσο του νέου ταμείου. Και αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αποκλείσουν αυτά τα προγράμματα από τον υπολογισμό του εθνικού χρέους και ελλείμματος. εφόσον οι εγγυήσει θα παρέχονται από την Ένωση. Οπότε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ε, συνάδελφοι, το νέο μας επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά μόνο την κινητοποίηση επιπλέον ε, χρηματοδότησης, αλλά και τον εντοπισμό των κατάλληλων προγραμμάτων και την παροχή της τεχνικής αρρωγής που χρειάζονται ώστε να, φτάσουν, να οριμάσουν γρήγορα. Αυτή θα είναι μια από τις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και δεν ανησυχώ για τα χρήματα, ανησυχώ για τα ε, προγράμματα, για τα σχέδια. Χρειάζεται εδώ να τα δουλέψουμε δηλαδή. Χρειάζεται να εντοπίσουμε αυτά τα προγράμματα ώστε να αντιστοιχούν στα τρία κεντρικά μας κύρια κριτήρια. Ε, καταρχήν, προγράμματα με σαφή προστιθέμενη, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δηλαδή που υποστηρίζουν τους ευρωπαϊκούς μας στόχους ε, όσον αφορά την ευφυή και καθαρή κινητικότητα. Και χτες είχαμε μια παρουσίαση για το νέο πακέτο διαχείρισης της ε, θαλάσσιας ναυσιπλοείας. Εξαιρετικό, συναρπαστικό έργο, ε, πολύ καλό παράδειγμα για το συνδυασμό των προσπαθειών των κρατών μελών. Ελπίζω πως θα έχουμε πολύ, πολλά περισσότερα τέτοιου είδους προγράμματα. Δεύτερο κριτήριο, ε, προγράμματα που να είναι οικονομικά βιώσιμα και με υψηλή κοινωνικο-οικονομική απόδοση που σημαίνει δουλειές. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα πραγματικά να ενθαρρύνω τους πάντες. Ας δημιουργήσουμε ευφυείς θέσεις εργασίας. Και γιατί, μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε ευφυείς θέσεις απασχόλησης είναι να βελτιώσουμε και έπειτα προγράμματα τα οποία να είναι αρκετά όρημα ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν το αργότερο εντός τριών ετών. Αυτό ήδη το ανέφερα προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια ε, τα οποία προσθέτουν ε, κοινωνικο-οικονομική απόδοση όπως είπαμε προηγουμένως και μπορούν να ξεκινήσουν εντός τριών ετών. Ο τομέα των μεταφορών μπορεί να ε, ε, προσφέρει τέτοιου είδου προγράμματα γιατί δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Επιταχύνουμε την διαδικασία απλά και ξεκαθαρίζουμε ε, την προετοιμασία. Ε, ο αριθμό των προγραμμάτων στον τομέα των μεταφορών στα επόμενα τρία χρόνια εκτιμάται σε πάνω από 100 δι ευρώ επενδύσεων. Λιμάνια, σιδηροδρομικέ γραμμές που οδηγούν σε αυτά, αναβάθμιση των καναλιών, αυτοκινητόδρομοι, αιτιές ε και τεχνολογίες καθαρών καυσίμων. Τα κράτη-μέλη έχουν δώσει στην Task Force Κομισιόν ΕΤΕΠ λίστες προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα τρία αυτά κριτήρια, εκ των οποίων μέγα τμήμα αφιερώνεται στις υποδομές των μεταφορών. Με την πρωτοβουλία, μετά από πρωτοβουλία της Αλκής Προεδρίας, η έκθεση Κριστόφερσεν που θα παρουσιαστεί αύριο στο Συμβούλιο Μεταφορών αυτή η έκθεση λοιπόν εντοπίζει προγράμματα για τους, τις μεταφορές, σε, ειδικά για τους διαδρόμους TNT, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο αυτό. Ήδη θα σας ενημερώσω για τα προγράμματα αυτά που έχουν εντοπιστεί από τον κύριο Κριστόφερσεν μαζί με τον Ευρωπαϊκό, Ευρωπαίο Συντονιστή Κάρλο Σέκη και Κούρτ Μπόντβιχ. Ορισμένοι διάδρομοι ε, καθώς ε, και κομμάτια που λείπουν από τις υποδομές, όπως ας πούμε η ε, σιδηροδρομική βαλτική σύνδεση ανάμεσα στη Βαρσοβία και το Ταλίν, καθώς και η οδική και σιδηροδρομική πρόσβαση στο λιμάνι της Βαρσελόνας η αναβάθμιση του καναλιού του Κίελου. Επίσης, διευκολυντές για τις επιχειρήσεις, όπως η ανάπτυξη των λιμανιών του Δουβλίνου και της Βαλέτα. Και στην τρίτη ομάδα έχουμε ε, προγράμματα αστικών μεταφορών, όπως ε, αυτό των Βρυξελών, το, η νέα γραμμή μετρό στο, στα πράσινα του Παρισιού ή υποδομές για την κινητικότητα με ηλεκτρισμό στο Τσεχική Δημοκρατία. Πολύ συγκεκριμένα προγράμματα από όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό σχέδιο αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία. Πρέπει να προσέξουμε ώστε οι ιδιωτικέ και οι δημόσιες επενδύσεις να υλοποιηθούν και αυτό θα γίνει αν μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον. Αυτή είναι η δουλειά μας. Για να προσελκύσουμε τους επενδυτές θα πρέπει να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι κανονισμοί θα είναι όσο γίνεται πιο απλοί και κατανοητοί, καθώς και να ε, ε, μεταρρυθμίσουμε τους πεπαλαιωμένους κανονισμούς. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ακριβείς οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις ε, αντικτύπου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρει εκκρεμεί πρωτοβουλίε για τι μεταφορέ στην παρουσίασή του την περασμένη Τετάρτη στο Κοινοβούλιο. Το τέταρτο σιδηρομικό πακέτο, τον ενιαίο ευρωπαϊκό ε, ε, ουρανό και την ε, πρωτοβουλία της γαλάζιας ζώνης. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι τεράστια σημασία ώστε ο τομέας των μεταφορών να καταστεί ελκυστικός για τους επενδυτές και αυτές αναφέρονται ως προτεραιότητες και στο δικό μου τη δική μου δήλωση της εντολής. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται για φακέλους που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο και ότι βρίσκονται και στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Μεταφορών αύριο, το τέταρτο συνδρομικό πακέτο, καθώς και το SES 2 sin αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να πιέσω το Συμβούλιο να ενεργήσει και να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μαζί σα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ελπίζω λοιπόν ότι εδώ θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, η θέσπιση του σωστού ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία μιας κατάλληλης πολιτικής για τις, για τις ε, υποδομές. Χρειάζεται να θέσουμε σε εφαρμογή την πρακτική ότι ο χρήστης πληρώνει και ο ρηπαίνων πληρώνει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα εισοδήματα από τις υποδομές θα επανεπενδύονται στις υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιοι από την Επιτροπή σας θα ήθελαν να δηλώσω κατά πόσο υποστηρίζω ή αντιτίθεμαι στο, στην γερμανική πρωτοβουλία ΜΑΟΤ. Θα το ξεκαθαρίσω αμέσως ε, στην γερμανική πρωτοβουλία για τα διόδια. Για το συγκεκριμένο θέμα, και θα το ξεκαθαρίσω αμέσω τώρα, και αντίθετα από τα προγράμματα χρέωσης για τα βαριά οχήματα υπό την οδηγία για την Ευρωβινιέτα, τα νομοσχέδια των κρατών μελών δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα, νομοσχέδια δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Οπότε η Κομισιόν θα έχει το δικαίωμα να λάβει επισήμω θέση για τη συμβατότητα των διοδίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα έχει οθετηθεί από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη φάση εγώ μπορώ μόνο να πω και να επαναλάβω κάποια βασικά στοιχεία. Ενώ η ε, Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή της αρχής ε, του «Ο χρήστης πληρώνει», θα προσέξει ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτό χρειάζεται να γίνει με τρόπο ώστε να γίνεται απόλυτα σεβαστές οι ευρωπαϊκές συνθήκες και οι αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτές των αρχών περί μη διακρίσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα συμβιβασμό από αυτού του σημείου και είμαι πεπισμένη ότι οι γερμανικές αρχές το κατανοούν απολύτως αυτό. Φυσικά και έδωσα οδηγίες στις υπηρεσίες της Επιτροπής να παραμείνουν σε στενή επαφή και να συνεργαστούν με τις γερμανικές αρχές ώστε να ε, τους παρέχουν ε, κάθε ε, συνεργασία. Και ίσως θα ακούσατε και στα νέα πως είχαμε μια πολύ θετική συνάντηση με το Γερμανό Αρμόδιο Υπουργό επί του θέματος. <clears throat> Όπως έχω προπεί λοιπόν, είμαι δεσμευμένη να συνεργαστώ μαζί σας στο πνεύμα αμοιβές κατανόησης και Σημειώνω την ψηφοφορία σας ε, σήμερα το πρωί. Φυσικά και ενημερωθήκαμε όσον αφορά την ε, ταξινόμηση των σοβαρών παραβάσεων στις οδικές μεταφορές που προτάθηκε από τον προκάτοχό μου τον κύριο Κάλλας. Μου είπαν ότι αυτό το κείμενο είναι αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων από τα κράτη-μέλη εδώ και δύο χρόνια σχεδόν και ότι η Κομισιόν έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια εντός του νομικού πλαισίου για την ώρα. Βεβαίως ε, είμαι έτοιμη να κοιτάξω ξανά αυτό το θέμα με για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αλλά ξέρετε ότι η βασική πρόκληση για την κοινωνική νομοθεσία δεν είναι η έλλειψη αυτής, αλλά περισσότερο η εφαρμογή της και η επιβολή των κανόνων που περιλαμβάνει. Περισσότερη νομοθεσία δηλαδή δεν σημαίνει καλύτερη πρακτική. Όπως θα θυμάστε, ήδη δεσμεύτηκα στη διάρκεια της ακρόασης να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα και να αποφύγουμε έτσι τις διαφορετικούς ορισμούς του, του κανονισμού. Γι' αυτό και είναι αρκετά εντυπωσιακό να βλέπω να απορρίπτεται μια πρόταση που αφορά καλύτερη εφαρμογή και κατηγοριοποίηση των ε, διαφόρων παραβάσεων. Μπορεί να είναι μόνο μια μερική λύση αυτή εδώ, συμφωνώ, αλλά τουλάχιστον είναι μια λύση που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό ίσως θα μπορούσατε να τη στηρίξετε. Φυσικά όμως σέβομαι τη γνώμη σας, όπως σέβομαι και τη ψήφο σας και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι πάντοτε υπάρχει χώρος για βελτίωση, για όλα. Οπότε σας καλώ να το έχουμε αυτό υπόψη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, Θέλω σύντομα να μπορέσουμε να εστιαστούμε στις νέες πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρθηκα στη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής σας ήδη. Θα ήθελα λοιπόν να συμβάλλω με αποφασιστικό τρόπο στις ε, προτεραιότητες τις οποίες εξέθεσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στις πολιτικές του κατευθυντήρης γραμμές. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι οι μεταφορές διευκολύνουν την ανάπτυξη, ότι έχουν μεγάλο δυναμικό όσον αφορά ε, την δημιουργία θέσεων απασχόληση και είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν μεταξύ τους οι περιφέρειές μας και να συμβάλλουμε έτσι ε, προς την μετακίνηση σε μια οικονομία που να είναι αποδοτική όσον αφορά την ενέργεια και ε, να καταναλώνει πολύ λίγο άνθρακα. Ε, διαρκώς λοιπόν θα έχω στο μυαλό μου και τους πελάτες μας, δηλαδή τους επιβάτες και τους ε, επιχειρηματίες και το να δημιουργήσουμε έτσι τις συνθήκες ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία των μεταφορών να ανθίσει. Ε, πιστεύω στεναρά στο ρόλο των τεχνικών και μη τεχνολογικών ε, καινοτομιών όπως καινοτόμα μοντέλα επιχειρηματικά, ως ένα παράδειγμα μη τεχνικής καινοτομίας, καθώς και τις καινοτόμες υπηρεσίες και πώς προς αυτό το σχέδιο για τις ευφυείς πόλεις θα είναι ένα από τα πρώτα στη δική μου ημερήσια διάταξη. Η Κομισιόν θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου και με χαρά θα μπορέσω να σας αναφέρω στους συντονιστές σας ε, τα σχετικά ήδη στη διάρκεια της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου. Απόψε θα συμμετέχω μαζί με τον κύριο Κράμερ σε μια ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους επιτρόπους και τους προέδρους των επιτροπών για αυτό το πρόγραμμα και με χαρά ε, περιμένω να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων ώστε να βοηθηθούμε να σχηματίσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2015 αλλά και γενικότερα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εδώ και ένα μήνα ε, έχω έρθει σε επαφή με πολλούς φορείς του τομέα των μεταφορών ώστε να μπορέσω να θεσπίσω συμπαγείς, στέρεες και καρποφόρες ε, σχέσεις συνεργασίας μαζί τους. Ε, θέλω να εξασφαλίσω ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί καλύτερα και γρηγορότερα προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού λαού. Επίσης σκοπεύω να κάνω τακτικές επισκέψεις στα κράτη-μέλη, ώστε να βλέπω συγκεκριμένα ποιος είναι ο αντίκτυπος των αποφάσεών μας, των αποφάσεων που λαμβάνουμε εδώ στις Βρυξέλλες, στις καθημερινές, πώς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και πώς τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε αναπτύσσονται. Και θα τολμήσω μάλιστα να σας καλέσω να έρθετε μαζί μου όταν θα επισκεφτώ τις χώρες σας ή και αλλού όταν θα πάω. Ελπίζω να εισακουστεί αυτή η ειλικρινής μου πρόσκληση για συνεργασία και πραγματικά προσβλέπω στην συνδημιουργία μιας δυναμικής, ενός δυναμικού και δραστήριου προγράμματος μεταφορών, σε συνεργασία μαζί σας. Ένα σύστημα μεταφορών το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί ως ένας αξιόπιστος μηχανισμός για, στον οποίο θα στηρίζεται επιτυχής ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ja, ευχαριστώ για την τοποθέτηση, για την πρόσκληση, για καλή συνεργασία. Νομίζω ότι και εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια καλή συνεργασία. Τόσο με την Επιτροπή όσο και με το Συμβούλιο, το αναφέρατε και εσείς ότι οι διαπραγματεύσει ε, για το τέταρτο πακέτο για οι σιδηροδρομικές μεταφορές κάπως έρνουν τα πόδια, αλλά πρέπει να προχωρήσουν για να προστατεύσουμε και το κλίμα και την οικονομία της Ευρώπης, τις μεταφορές της Ευρώπης και τις θέσεις εργασία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά για την τοποθέτηση σας και πάλι ευχαριστούμε που ήρθατε και ακούμε στον πρώτο γύρο τους συντονιστές. Έχουμε ένα κάποιο περιορισμό χρόνου με δύο λεπτά μόνο για τους συντονιστές που θα τους ακούσετε όλους για να απαντήσετε στη συνέχεια και μετά τους λοιπούς συναδέλφους που θα έχουν ο καθένας από ένα λεπτό και πάλι αφού τους ακούσετε θα μπορέσετε να απαντήσετε. Αν είμαστε όλοι προσεκτικοί με το χρόνο θα, μπορέσετε, θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Φαντακάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να σας καλωσορίσω κυρία Μπούλτς. Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μαζί σας, εμείς από την Επιτροπή Μεταφορών. Βλέπετε ότι η αίθουσα είναι γεμάτη. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που έχουμε για τη δική σας εργασία. Ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε και να κάνουμε επικοδομητική κριτική. Δύο λεπτά έχω μόνο στη διάθεσή μου και γι' αυτό και θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα επενδύσεων του κύριου Γιούγκερ και την ευελιξία του. Πόσο ευέλικτο είναι αυτό το πρόγραμμα τελικά. Υπάρχουν ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν, ιδιωτικές εταιρείες μεγάλες. Θέλει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και Υπάρχει φόβος ότι θα υπάρξει απώλεια επιδοτήσεων και ενισχύσεων με την έλευση του ιδιωτικού τομέα. Μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Δεύτερον, ο πρόεδρος Γιούνκερ συνεχώς λέει ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να επενδύσουν. Ωστόσο, τα ποσά και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ υψηλά. Από την άλλη πλευρά, κανείς στην Ευρώπη δεν περιμένει ούτε ελπίζει σε ένα ενιαίο σύστημα διοδίων. Όμως, με τη νέα τεχνολογία, με αυτά τα ενοποιημένα συστήματα, ελπίζουμε να, η ίσπραξη των διοδίων να είναι πολύ πιο εύκολη. Μπορεί να γίνει αυτό με πιο απλό τρόπο και ελπίζω ότι θα κάνετε το παν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί τελικά θα ήταν κρίμα να βάλετε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναλάβουν αυτό το φόρτο, να συμμετάσχουν και τελικά να τους πείτε ότι δεν θα εγκρίνετε τα σχέδιά τους και τα έργα τους. Μπορείτε επίσης να μας πείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό τα επόμενα χρόνια γιατί θέλουμε η βιομηχανία μεταφορών πραγματικά να μπορέσει να επιβιώσει. Ευχαριστώ κύριο Σερτού. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε και εμείς από τους δονηστές. Σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας στην επόμενη πενταετία. Θα σας παρακολουθούμε, θα σας συνοδεύουμε σε αυτό το έργο. Τρεις ερωτήσεις έχω προς εσάς κύριε Επίτροπε. Καταρχάς για να επανέλθω και στο πιο δυσάρεστο για σας, το θέμα του, ε, των διοδίων από πλευρά τη Γερμανία. Από χθε λοιπόν ακούστηκε από το Υπουργείο των Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανία ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία λέει ότι σε ορατό μέλλον θα επιβαρυνθούν σημαντικά και οι Γερμανοί οδηγοί των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ε, οχημάτων στη Γερμανία με αυτό το τέλος διοδίων. Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να το δεχθείτε. Βέβαια πρέπει να σας ρωτήσω το εξής, γιατί φαίνεται ήδη να παγιώνεται η εικόνα ότι η Γερμανία προσπαθεί να εισαγάγει δύο διαφορετικούς νόμους, χωριστούς. Έναν που θα είναι προς τα έξω ορατός, για να είναι αποδεκτός με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ένα εσωτερικό, ο οποίος θα κάνει την διαφοροποίηση και θα μειώνει την επιβάρυνση για το γερμανό οδηγό. Εσείς λοιπόν βλέπετε να είναι αυτό συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και δεύτερον, στα κοινωνικά ζητήματα. Ε, λέτε στην δήλωσή σας της τέταρτη σελίδα, εν της ακροάσεως, ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμήσετε το κοινωνικό dumping. Τι συγκεκριμένε προτάσει έχετε να μας φέρετε σήμερα για το θέμα αυτό. Τρίτη ερώτηση, το σχέδιο 10 σημείων της ε, Επιτροπής Juncker και του Πρόεδρου Juncker δεν αναφέρει πουθενά το χώρο των μεταφορών. Τι σημασία έχει λοιπόν για την Επιτροπή Juncker ο τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ, Ρόμπερτ Σίλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, καλωσορίσω εκ μέρους του, της πολιτικής ομάδας του ECR. Έχουμε τα χρήματα, έχουμε τα αξιόπιστα έργα και τις σωστές επενδύσεις. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες. Ωστόσο, με ανησυχεί όλη αυτή η εξέλιξη. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στο συνδέοντας την Ευρώπη έτσι ώστε όλα τα project για όλους τους διαδρόμους να είναι τα καλά και να συνδέσουν περιοχές χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Το σημαντικό είναι τι νομίζει η αγορά για όλα αυτά. Στα ηθορία είναι πολύ καλά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Οι χρήστες πληρώνουν, ο πληρώνουν, τα χρήματα από τις επενδύσεις ε, μένουν στον τόπο εκεί που, που προέρχονται. Ωστόσο, Θα πρέπει να δοθούν κονδύλια για μεγάλα project υποδομών, δελειώς όλο και περισσότερες περιοχές θα ε, δουν τον πληθυσμό τους να τις εγκαταλείπει. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι κάπως περίπλοκη η κατάσταση που περιγράφεται. Βάζετε 10% των χρημάτων σε ένα νέο ταμείο και αυτό είναι ρίσκο. Υπάρχει ένα κατόφλι ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, π.χ. τα 10 που θα μπουν στο project συνδέοντας την Ευρώπη. Αν το 85% είναι συγχρηματοδότηση με εσά, το 15% θα έρθει από το νέο ταμείο και οι τοπικές αρχές δεν θα εμπλακούν καθόλου. Έχετε απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικό για μας τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ στα θέματα κοινωνικού ντάμπιν και εργασιακού ντάμπιν μάλλον, αλλά θα επανέλθω αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την τοποθέτησή σας, την αναγγελία των σχεδίων σας. Νομίζω ότι θα ανακαλύψει κατά στιγμή ο κύριος Γιούνκερ ότι χωρίς μεταφορές δεν υπάρχει τίποτα. Ε, βλέπουμε τις μεταφορές πάντοτε όσο το σύστημα κυκλοφορίας του αίματος, κυκλοφορικό δηλαδή και όχι κυκλοφοριακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς μεταφορές δεν υπάρχει. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει εσωτερική αγορά. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη η Επιτροπή Γιονκέρ. Και επίσης για τις επενδύσεις, το πακέτο με τις επενδύσεις και τις δυνατότητες για καλύτερη χρηματοδότηση. Ε, είπατε εσείς ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί να επενδύσουν τίποτα τα κρατημέλη. Τουλάχιστον εγώ αυτό αντελήφθηνα από τα λόγια σα, ότι δηλαδή μπορούν να διαγράψουν, να αποκλείσουν από το χρέο του τα έργα, τα επενδυτικά και ότι μπορεί να προσελκύσουν θετικά κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσει θα στραφούν κυρίω στις οδικέ μεταφορέ στην κατασκευή δρόμων, γιατί βλέπουμε ότι η τάση είναι αυτή και ίσω να χαθεί εκεί πέρα η πρόβλεψη για του υδροδρόμους για το θέμα των διοδίων. Ξέρω, ξέρετε ότι έχω καταθέσει και ερώτηση για το αν είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Από την άλλη, έχω όμως πληρωματικές ερωτήσεις. Η αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει και μένα ουσιοδέστατη. Εάν λοιπόν μου πείτε ότι δεν πρέπει να πληρώνει κανείς διόδια για τα ε, οχήματα με κινητήρα και μόνο ανάλογα με την χρήση πληρώνει κανείς το τέλος ή την επιβάρυνση, σε σχέση με το περιβάλλον, του, θα συμφωνήσω απολύτω. Κάτι ακόμη, ε, ζητήσατε την υποστήριξή μας, ε, την παρουσία μας, τις επισκέψεις στα κράτη-μέλη. Εάν υπάρχει δυνατότητα και ο χρόνος πολύ ευχαριστώ. εγώ θα είμαι παρούσα εάν μου το ζητήσετε για τη Γερμανία, αρκεί να μας λέτε και να μας ενημερώνετε και πού είναι τα πιο εντό εγωγικών διστακτικά κράτη, ώστε να ερχόμαστε και εμείς και να ενισχύουμε τις τάξεις σας με περισσότερη πίεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επίτροπο κυρία Μπούλτς και εγώ προσμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστούμε με εσάς, με όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και με ε, τις χώρες μέλη. Με χαρά παρακολούθησα τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών να είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη, να παρουσιάζει μεγαλύτερη συνέπεια. Όσο εκ τούτου, Ερωτώ, τι είδου στήριξη περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δική σας δουλειά, πώς μπορούμε να σας στηρίξουμε. Πράγματι, και εγώ επιθυμώ το σύστημα μεταφορών μας να, είναι πιο, να λειτουργεί πιο εύρυθμα, να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον υπάρχει, είναι πολλές οι προκλήσεις σε σχέση με την ενέργεια που προέρχεται από τον άνθρακα, σε σχέση με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας, θα τα αντιμετωπίσουμε πιστεύω ότι κρύβουμε τα μεγάλα προβλήματα. Δεν προχωρούμε αρκετά γρήγορα. Και αργά ή γρήγορα μετά την Παγκόσμια Συμφωνία για το Κλίμα, το σημείο εστίασης από την ενέργεια και το, τη βιομηχανία θα στραφεί πλέον στις μεταφορές, οι οποίες είναι ένας κλάδος που πραγματικά ε, δημιουργεί και αυτός ε, μόλις η ρήπανση. Επομένως υπάρχουν ευκαιρίες, μπορούμε να έχουμε πιο διαφανή, πιο πράσινη πολιτική μεταφορών, η οποία θα δημιουργήσει καλύτερο περιβάλλον στις πόλεις και θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πώς μπορούμε λοιπόν να δράξουμε αυτή την ευκαιρία, να λειτουργήσουμε πιο ενεργητικά, πιο δραστικά αν θέλετε. Θα είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα δώσετε προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρυμαντελή. Ευχαριστώ η κυρία Κα... Καλωσορίσατε, καλημέρα. Ε, ορίσατε κυρία Επίτροπε στην ε, Επιτροπή μας, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα να σας απευθύνω. Γρήγορα, σε πρώτη φάση, τι θα κάνετε για να ενοποιήσετε τις ε, πολιτικές μεταφορών εν ώψη της διάσκεψης για το κλίμα. Είμαστε στην κόπ της Λίμα του Περού. Και στη συνέχεια θα έχουμε το Παρίσι, όπως γνωρίζετε. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε ρόλο να διαδραματίσετε σε αυτή την κόπτη διάσκεψη για το κλίμα την προπαρασκευαστική, όπως και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα άμεσα, γιατί ο κλάδος των μεταφορών εξαρτάται ιδιαίτερως από το ε, πετρέλαιο και έχουμε και όλες τις κλιματικές αλλαγές και τις σύγχρονες, σύγχρονες τάσεις που θέλουν τη μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, σχέδιο αστικής κινητικότητας είναι προτεραιότητα. Ε, οι μετακινήσεις στο άστι. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να μας, παρουσιάσετε, να μας και δεν μιλήσατε καθόλου για την αεροπλοεία η οποία είναι ένας κλάδος που εκπέμπει εξαιρετικά υψηλά, σε εξαιρετικά υψηλές ποσότητες αέρια που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το καθεξής. Και το θέμα του ντίζελ είναι στις προτεραιότητές σας, γιατί μιλούμε για μεγάλη μόλυνση και ρήπανση σήμερα. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο 300 δις. Ωστόσο, πώς μπορεί να εγκρίνει σχέδια άχρηστα. Λέτε εσείς ότι θέλετε να εγκρίνετε σχέδια που θα είναι οικονομικώς ε, βιώσιμα. Όμως, έχετε εγκρίνει σχέδια όπως αυτό που ενώνει τη Λιόν με το, με το Τωρίνο, όπου η απόδοση επί της επένδυσης πραγματικά δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Έχουμε το, το θόρυβο, τα επίπεδα θορύβου, τα ατυχήματα. Όλα αυτά τα έχετε λάβει υπόψη σας. Σήμερα δεν νομίζω ότι υφίσταται αυτή η αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κυρία Μπούλς. Δεν ήθελα καταρχάς να πω ότι βλέπουμε να υπάρχουν πράγματα που, όπου δεν λειτουργεί σωστά η ίδια η νομοθεσία. Το καμποτάζ, οι μεταφράσεις, μεταφορές μικρών υποστάσεων στα εσωτερικά ύδατα δεν λειτουργούν καλά. Βλέπουμε στην Σουηδία το πρόβλημα της ε, μεταφοράς ε, μεγάλων φορτίων που πρέπει να περάσουν από την Δανία και μετά να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην Σουηδία. Εσωτερικές μεταφορές που ουσιαστικά δεν, δεν αξίζουν οικονομικά, δεν είναι οικονομικά συμφέρουσες. Και έχουμε επίσης τους οδηγούς αυτούς οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες με 500 ευρώ το μήνα να οδηγούν καθημερινά χωρίς ανάπαυση, να ε, τρέχουν από τη μια άκρη της Ευρώπης μέχρι την άλλη. Τρώνε τίποτα λαχανικά στο δρόμο, δεν έχουν ούτε ντους να πληθούν. Σκανδαλώδεις συνθήκες ε, που προξενεί αυτός ο κανονισμός του Καμποτάζ και που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί δίνεται πολύ λάθος εικόνα και επίσης έχουμε και πλαστές άδειες οδήγησης. Στη Σουηδία ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι εύκολο να αγοράσει κανείς για μερικές εκατοντάδες ευρώ άδεια οδήγησης μέσω του ίντερνετ, γιατί είναι δύσκολες εξετάσεις οι κανονικές, με 300-400 ευρώ μπορεί κανείς να αγοράσει μέσω ίντερνετ και έχουμε οδηγούς που δεν ξέρουν καν να οδηγούν ε, φορτηγά οχήματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, Και τώρα κλείνω... Αυτό ήταν ο πρώτο γύρο ε, με του συντονιστέ. Κλείνω τον κατάλογο τώρα. Οι επόμενοι ομιλητέ θα έχουν από ένα λεπτό, αλλά καλώ την Επίτροπο να δώσει απαντήσει. Ευχαριστώ τους ε, κυρίους και κυρίες βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Με χαροποιεί το γεγονός ότι έχετε τόσο πολύ ενδιαφέρον ε, για τα θέματα αυτά. Αυτό άλλωστε είπα και στο τέλος της ομιλίας μου ότι θα είναι οι μεταφορές, ο κύριος κινητήριος μοχλός, ε, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας και πάνω απ' όλα αυτή που θα δημιουργήσει και θέσει εργασίας. Άρα πρέπει να την υποστηρίξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη πενταετία. Τώρα για να απαντήσω στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς σας. Ο συνάδελφός μου εδώ με βοηθάει και τον ευχαριστώ γιατί μου, με βοηθάει ακόμα και να ε, σημειώσω, να κρατήσω τις σημειώσεις των ερωτήσεών σας. Εάν τυχόν κάτι ξέχασα βεβαίως θα επανέλθω με κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Μία-δύο αναφορές στο πακέτο αυτό των μέτρων για 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Κάμπ ε, έθιξε το σύντημα πρώτος, αλλά και κάποιοι άλλοι βουλευτές. Αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι αυτά τα 300 δις, 315 δις, δεν είναι χρήμα που θα στερηθεί κάποιο άλλο έργο ή πρόγραμμα. Είναι ένας μηχανισμός. Παίρνουμε 10% από τα έργα ΣΕΦ για να έχουμε τη μόχλευση και θα μας δώσει 100 δις σε επενδύσεις δυνητικά. Μόνο όμως για έργα τα οποία είναι όριμα η δική μας η εκτίμηση είναι ότι στην κοινότητα ΣΕΦ υπάρχουν επαρκώς, υπάρχει επαρκής αριθμός, επαρκώς ορίμων έργων για να χρηματοδοτηθούν με το μηχανισμό αυτό, αλλά βέβαια αρκετή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμη. Οι μεταφορές πιστεύω ότι θα επωφεληθούν τα μέγιστα, διότι θα είμαστε δικαιούχοι για το 1 τρίτο περίπου του συνολικού προϋπολογισμού αυτού του ταμείου. Άρα μπορεί εσείς να αναφέρεστε ότι η ε, το πρόγραμμα ή τα σημεία Juncker δεν αναφέρουν ρητά τις μεταφορές. Είμαστε παρόντες παντού και στη θέση εργασίας και στη δημιουργία ανάπτυξης και στο, στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου. Όπου και να κινηθεί κανείς βλέπει τις μεταφορές ως καθοριστικό στοιχείο. Ίσως θα έπρεπε ρητά να αναφερθούν. Θα κοιτάξω μήπως και καταφέρω να φέρω κάποια ε, αλλαγή. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση στο θέμα αυτό και αν κοιτάξετε το Twitter και το Facebook, τους λογαριασμούς μας, θα δείτε ότι είμαστε και η πιο δραστήρια ομάδα. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε για το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, τι ωφέλη προκύπτουν από τις δράσεις μας. Και όταν λέω μας, ενώ όλων ημών που εμπλεκόμεθα στις μεταφορές, γιατί ό,τι αποτέλεσμα έχουμε προκύπτει από την κοινή μας δουλειά. Είχα εδώ κάτι άλλο συγκεκριμένο για τις μεταφορές. Ξέρετε ότι στους επόμενους μήνες ε, έχουμε κρίσιμη περίοδο για αυτά τα 315 δις. Προσπαθούμε και θα βγούμε εξ προς τα έξω να κερδίσουμε την υποστήριξη του κοινού, να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, να καταστούμε ελκυστικοί για τους επενδυτές. Είναι μια δουλειά που μόλις αρχίζει. Ελπίζω όμως με τη δική σας βοήθεια και με τη δική σας βοήθεια να πάει καλά. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι, γιατί με ρώτησε και ο κύριος Ζήλε κάτι σχετικό, ότι υπάρχουν και διαφορετικοί μηχανισμοί, το Ταμείο Συνοχής, παράδειγμα, τα Ταμεία Συνοχής, αλλά παραμένουν αλόβητα, δεν περιορίζονται σε τίποτα. Δεν τους στερούμε τίποτα. Έχουμε το μηχανισμό 240 με τεράστια ποσά για τις υποδομές από τα οποία τα περισσότερα θα είναι έργα υποδομών. Συγκεκριμένα νούμερα δεν έχω να σας πω για τη Σλοβενία, όμως έχουμε 1,2 δις για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και τα περισσότερα, όπως είπα, από τα κονδύλια πάνε στις μεταφορές. Αυτός είναι ένας μηχανισμός. Ο άλλος είναι αυτός του παραδοσιακού δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξακολουθεί να λειτουργεί. Μετά μπορεί να έχετε ακούσει ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός καινούριο για τα μακροπρόθεσμα έργα, ε, επενδυτικά έργα. Και θα ξεκινήσει και αυτός. Διαφορετικοί λοιπόν μηχανισμοί για διαφορετικού τύπου έργων, για διαφορετικών τύπων έργα και αυτός ο πρόσθετος μηχανισμός θα είναι διαθέσιμος για τα έργα που είναι όριμα, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν να λειτουργούν σε δύο έργα που θα έχουν κοινωνικο-οικονομικό ε, αντίκτυπο, αλλά βέβαια θα χρειαστούν ε, επενδυτές. Πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και να προσελκύσουμε τους επενδυτές. Δεν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν αυτόματα. Δεν θα ξεκινήσει αυτός ο μηχανισμός να λειτουργεί αυτόματα. Ναι, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να καθυστερώ πολύ για το ένα μόνο θέμα. Μετά υπήρξε ένα θέμα για τις αεροπορικές μεταφορές και τον ανταγωνισμό. Έχει ξεκινήσει διάλογο η Επιτροπή στον τομέα αυτό με τις περιφέρειες. Είχα υπόψη μου εγώ τις αεροπορικές εταιρείε του Περσικού υπεραδειγματικού Όλπου. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό το διάλογο με ε, σκοπό να ενισχύσουμε και τη διαφάνεια και τις ασφαλιστικές δικλίδες για να εξασφαλίσουμε και θεμητό ανταγωνισμό. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση του διαλόγου τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες η πλευρά του Περσικού κόλπου δεσμεύθηκε για βήματα προς θεμητό ανταγωνισμό. Μικρά βήματα, αλλά ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε τις επραγματεύσεις και τις συνομιλίες. Και από κοινού συντάκτηκε ένας οδικός χάρτης με τη σύνταξη μιας ομάδας που θα παρακολουθεί και την υλοποίηση. Ο προσεχής ε, διάλογος αναμένεται να αναπτυχθεί στο Κατάρ το Μάρτιο του 2015. Όπως είπα ξεκινάμε τώρα. Έχουμε τα θέματα των ανοιχτών ουρανών, των ανοιχτών εθέρων και έχουμε και άλλα θέματα σχέση με τη Ρωσία, και ζητήματα από τα οποία εξαρτώ, για τα οποία εξαρτώμεθα από τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι με το που θα βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση, θα ανασκουμποθούμε και θα προσπαθήσουμε και για τις ενέργειες μεταφορές για τον ενέργειο χώρο να εξασφαλίσουμε συμφωνία. Ο κύριος Ερτού μου έθεσε μια σειρά ερωτήσεων, ελπίζω να μπορούσα να τις καλύψω όλες. Η μία αφορά το, την αποσύνδεση του συστήματος της βινιέτας ε, με τη φορολογία ή του, των διοδίων. Κοιτάξτε, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω για το θέμα αυτό και ζητώ την κατανόησή σας, γιατί δεν έχω δει τίποτα επί χάρτου. Τα πάντα είναι φήμες, τι υπόθηκε, τι σχολιάστηκε, τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Τον Υπουργό ρώτησα και μου εξήγησε κάποια πράγματα, αλλά αναγκάστηκα να του πω άστο, άστε να το δω όταν θα είναι έτοιμο. Άρα η μόνη θέση που μπορώ προς το παρόν να υιοθετήσω είναι no comment, ουδέν σχόλιον, μέχρι να είναι έτοιμα οι προτάσεις επί χάρτου, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Παρακολουθούμε πάντως εκ του σύνεγγης. Έγινε. Έγιναν συνομιλίες άτυπες με τους ε, Γερμανούς εταίρους και συναδέλφους. Ε, τους προσφέραμε κάθε υποστήριξη και αρρωγή ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για προσφυγή στη δικαιοσύνη, η ανάληψη μάλλον ε, ενόμων μέτρων, ε, αλλά βέβαια είμαστε και θεματοφύλακα των συνθήκων και ως εκ τούτου εάν μας συμβουλεύσουν σχετικά οι νομικές υπηρεσίες, πάνω σε αυτές θα στηριχτώ, θα πάρω καμιά απόφαση με τη δική μου προσωπική κρίση, θα αναλάβω δράση και δικαστική. Τέλος ο χρόνος μου! Όχι, λέει ο πρόεδρο. αλλά σας διακόπτω γιατί εάν μιλάτε τόσο πολύ θα πρέπει να μείνετε παραπάνω χρόνια. Έχουμε ακόμα 25 ερωτήσεις που πρέπει να λάβουν απαντήσεις. Καλώς, λέει κυρία Μπούλ. τότε πολύ σύντομα να πω δύο λόγια για τα ζητήματα τα οικολογικά. Ε, είμαι αφοσιωμένη στην, ε, στο πράσινο, στην πράσινη ατζέντα, στο πράσινο θεματολόγιο. Ε, το θέμα της ε, αξιοποίησης ε, πετρελαϊκών πόρων κατά 93% ως ενέργεια στην Ευρώπη με συγκλώνησε όταν το είδα. Τα ποσοστά είναι, συντριπτικά και πρέπει να μειωθούν σημαντικά και αναλόγως θα μειωθούν και οι εκπομπές του οξυδιού του άνθρακα. Συμφωνώ με την κυρία Βουλευτή που το ανέφερε. Ωστόσο, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω και να προδικάσω θέσεις που θα παρουσιαστούν μετά τα Χριστούγεννα, σας διαβεβαιώνω ότι μόλις είναι έτοιμες θα έρθουμε να σας τις ε, εξηγήσουμε και ελπίζουμε να εξασφαλίσουμε και την υποστήριξή σας. Επίσης, μια-δυο ερωτήσεις αφορούσαν το εξωτερικό κόστος, το οποίο θέλουμε να ενσωματώνεται στις ε, λογιστικές καταγραφές των μεταφορών και τους μηχανισμούς χρέωσης. Ενδείξεις υπάρχουν από ευρωπαϊκά κράτη ότι ήδη το πράττουν. Άρα εμείς ε, ενθαρρύνουμε και παρακολουθούμε τις, ε, τους απολογισμούς αυτούς και, τις, και συνοδεύουμε τις επιλογές Άρα θέλουμε συμπερίληψη του εξωτερικού κόστους στο όλο κόστος. Η κυρία Ντέλη επίσης αναφέρθηκε σε δράσεις για το COP15. Αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες ε, του Αντιπρόεδρου Σεφτσοβιτς. Σας το λέω εξ αλλά και εμείς θα διαδραματίσουμε το ρόλο μας και θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά τα Χριστούγεννα για τις θέσεις μας, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξή σας και να προχωρήσουμε με κοινή συνεννόηση σε άτυπες συνομιλίες. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω στα σχόλια των στις ερωτήσεις μάλλον των συναδέλφων για, τις, για τους επενδυτές από τρίτες χώρες. Ευπρόσδεκτη είναι, αυτό θα σας πω. Ας έρθουν να επενδύσουν στις υποδομές για και το πού και πώς τους όρους, τις προϋποθέσεις θα τους προσδιορίσουμε ακόμα. Αλλά πάντως από τα τελευταία στοιχεία που έχουμε βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε περίπου 700 δις ευρώ εν όλο για να εξυγχρονιστούν οι μεταφορές. Και αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα πολύ κακών επιλογών και συμπεριφορών στο παρελθόν. Τώρα εμείς πρέπει να πληρώσουμε τα σπασμένα και αναγκαστικά θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδυτές. Μόνοι μας δεν τα καταφέρνουμε. Ο κύριος Λούντκρεν, αλλά νομίζω και η κυρία και ο κύριος Ερτού με ρώτησαν ε, για κοινωνικό ντάμπινγκ και τα σχετικά συστήματα. Εμένα σε αυτά που σας είχα πει και στην ακρόασή μου το κοινωνικό ντάμπινγκ και η κατ' ουσίαν εκμετάλλευση της δουλειάς των ε, οδηγών, ο αθέμητος ανταγωνισμός, πάντα, όπως σας είπα, λαμβάνει και στην ακρόαση λαμβάνει χώρα στο όριο των νόμιμων μεταφορών. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα βέβαια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο όπου υπάρχει πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό. Πρέπει να αξιοποιείται το κανονιστικό πλαίσιο. Η συμμόρφωση έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά συμμόρφωση σημαίνει ευθύνε για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα των μεταφορών και όχι μόνο για την Επιτροπή. Η υλοποίηση, ξέρετε και η εφαρμογή, είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εδώ ζητώ τη βοήθειά σας. Βοηθήστε με να εξασφαλίσω ότι τα κράτη-μέλη πράγματι θα ενστερνιστούν αυτούς τους κανόνες. Ζητώ τη βοήθεια σας γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και πάντοτε βέβαια θα προάγω την ε, νοοτροπία και την αντίληψη της συμμόρφωσης και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώσω τα αποτελέσματα. Ναι, Πρόεδρε, ξέρω, ήθελα να απαντήσω σε κάθε τι στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Καλώς λέει ο πρόεδρος γιατί έχουμε μόνο 25 ακόμα ερωτήσεις. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ λέει ο πρόεδρος. Καλώς ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, κάποια σχόλια ήθελα να κάνω. Δεν θα έχουμε καλή αγορά μέχρι ότου παραμεριστούν τα διάφορα συμφέροντα, τα εμπλεκόμενα οι επενδυτές πρέπει να πιστέψουν ότι γίνεται σωστή διαχείριση των project για να μπορέσουν να επενδύσουν. Το θέμα είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δουλειά του Επιτρόπου Μεταφορών και της Επιτροπής Μεταφορών είναι οι μεταφορές, όχι τόσο το περιβάλλον ή τα άλλα ζητήματα. Βεβαίω και αυτά είναι σημαντικά και τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι ο πυρήνα της δουλειά μας. Αυτά υπάρχει Επιτροπή Περιβάλλοντος να ασχολείται με αυτά, για παράδειγμα. Να συμφωνήσω με τα σχόλια του κυρίου Ζήλερ για τις λεπτομέρειες αυτής της χρηματοδότησης. Ωστόσο εκφράζω την απογοήτευσή μου. Εγώ έρχομαι από ένα νησί και το 84% των ανθρώπων που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχονται πετώντας με πτήσεις και το Ηνωμένο Βασίλειο συμβάλλει ιδιαιτέρως ε, τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι το ΣΕΣΑΡ, η αεροπλοεία και όλα αυτά δεν αναφέρονται επαρκώς. Είναι πολύ σημαντικές υποδομές, πολύ μεγάλες. Καλό θα είναι την επόμενη φορά που θα έρθετε να μας επισκεφτείτε να τα τονίσετε περισσότερο αυτά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ, Λουίς Δεκράντες Πασκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στον πραγματικό κόσμο, αγαπητή κυρία Επίτροπε. Στην ακρόαση αναγκαστικά, αν μιλήσαμε γενικώ, τώρα μιλούμε πολύ, ε, επί πολύ συγκεκριμένων πραγμάτων. Όλοι αυτό κάνουν και εγώ το ίδιο κάνω. Η Ισπανία λοιπόν ελπίζει πολλά με ε, το σχέδιο Juncker. Θα πρέπει να συμβάλλουν οι μεγάλες χώρες. Έχουμε τα όρημα έργα με αυξημένη προστιθέμενη αξία και σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Η Ισπανία θέλει να ξεφύγει πλέον από αυτή τη μέγενη της ανεργίας ε, συγκεκριμένα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις που μόλις τώρα ανέφερα και που είναι απαραίτητα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτά. Και το σχέδιο Juncker, ξέρετε, ε, ε, δεν περιλαμβάνει έχει κάτι το πολύ σημαντικό. Η συνεισφορά των κρατών μιλών για την υλοποίηση του project δεν θα καταλογίζεται ως μέρος του ελλείμματος και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε επιτέλους να ξεφύγουμε προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Κύριος Πέτερ Φαντάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι θα πρέπει την επόμενη φορά που θα έρθετε να έχουμε προβλέψει περισσότερο χρόνο στην ημερήσια διάταξη για τη συνάντηση μαζί σας, γιατί και είναι δύσκολο να ε, προλάβουμε να τα πούμε όλα, και εμείς και εσείς. Προτείνω λοιπόν να παραμείνετε στο θέμα των eco των πολύ μεγάλων φορτηγών για να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και δεν μιλήσατε καθόλου για το κοινωνικό ντάμπινγκ και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μπει στην κορυφή του καταλόγου των προτεραιοτήτων σας. Είμαστε σε οικονομικά χαλεπούς καιρούς και... Καλό θα είναι αυτό να είναι η προτεραιότητά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζώσπαχ. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχουμε διαπιστώσει νομίζω μια νέα δυναμική και έναν τρόπο για, τους, για τις μεταφορές και χαίρομαι ιδιαίτερως. Θα ήθελα να φερθώ λοιπόν τώρα στις οδικές μεταφορές όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα το κοινωνικό ντάμπινγκ στο οποίο αναφερθήκατε προβλήματα που έχουν να κάνουν ε, όχι μόνο με τους οδηγούς αλλά και με τεχνικές ελλείψεις και θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι θα πρέπει να, αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να συνδυαστούν όλα αυτά τα πράγματα σε έναν φορέα, ίσως όχι υπηρεσία ακριβώς, αλλά έναν φορέα που θα μπορεί να τα διαχειρίζεται όλα αυτά. Στο θέμα των μεταφορών διαπιστώνουμε προβλήματα όχι μόνο ως προς, τις, ε, ε, ως προς τα κάψιμα που χρησιμοποιούνται αλλά και ως προς την ε, χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ευχαριστώ πολύ, Κριστίνα. Merci, Madame la Commissaire. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσίασή σας και για αυτές τις πρώτες απαντήσεις σας, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Θα επανέλθω επί τριών σημείων της παρέμβασής σας. Πρώτον, το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Μας μιλήσατε με αισιόδοξο τόνο και θεωρείτε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Εάν όμως δεν έχει προχωρήσει το πολιτικό σκέλος μέχρι το καλοκαίρι της συμφωνίας αυτή, τι θα κάνετε για το τεχνικό σκέλος, το οποίο πράγματι έχει προχωρήσει αρκετά. Και είναι ένα ερώτημα που έχω θέσει και στον προκάτοχό αυτό καταρχάς. Δεύτερον, για τις επενδύσεις στις μεταφορές και το σχέδιο Juncker. Να σας πω ότι δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένη, διότι σας άκουσα να λέτε ότι πιστεύετε ότι θα αποκλείσετε από τον υπολογισμό του χρέους τη συμμετοχή των κρατών μελών. Αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό, όμως για ποια ποσά μιλούμε πριν φτάσουμε στα 100 δις, από τη στιγμή που καλυφθούν τα 100 δις προβλέπεται αυτή η ρύθμιση. Υπάρχει ένας ελάχιστος κύκλος αρκετά ενδιαφέρον. Το τρίτο ερώτημα δεν έχω χρόνο να το θέσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την Επίτροπο. Μια-δύο ερωτήσεις ε, γίνεται για, λόγος για τον οδικό χάρτη, υπάρχει ήδη αυτή η ιδέα για τα προγράμματα. Θα ήθελα να γνωρίζω κάποια πράγματα περισσότερα για τον τρόπο επιλογής, δηλαδή αυτή η, επιλογή, αυτή η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, καθώς και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για να τεθούν σε εφαρμογή τα προγράμματα αυτά. Και δεύτερον, ε, μια ερώτηση για το καμποτάζ, γιατί το υπογράμμισαν πολύ την ανάγκη μιας επίγουσας ε, παρέμβασης καθώς ε, οι αρνητικές επιπτώσεις φαίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό διερωτάμε μήπως υπάρχει κάποια μελέτη, αν γίνεται μελέτη ή αν πρόκειται να γίνει μελέτη, για να επαληθεύσουμε τις πρακτικές ε, επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια πρόταση τροποποίησης όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Μασιμιλιάνο Σαλίνη, ευχαριστώ. Ε, καλωσορίσατε κυρία Επίτροπε και εύχομαι ε, καλή επιτυχία. Κάτι για το CEF, η σχέση μεταξύ του CEF και του νέου προγράμματος επενδύσεων που πρότεινε ο Juncker. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. 3,3 δις, από όσο γνωρίζουμε, θα είναι το τμήμα της συμβολής του CEF στο νέο ταμείο. Οπότε είναι ξεκάθαρο το πώς θα, πώς ε, βρίσκουμε τα 16 δις της συμμετοχής στο Ταμείο. 3,3 είναι ένα καλό ποσό, απλώς ε, δεν θα ήθελα να βγουν κι άλλα από το, από Και η πρώτη μου σκέψη είναι η εξής όλες οι επενδύσεις δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό αποζημίωσης. Οπότε το να αφαιρεθούν 3,3 από το ΣΥΕΦΗ να μπουν στο πλάνο και ελπίζοντας ότι θα μοχλεύσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, σημαίνει επενδύσεις με γρήγορη ανταπόκριση και ανταπόδοση. Αυτό δεν είναι βέβαιο. Σίγουρα από δική μου πείρα για τις δικές μου επενδύσεις ξέρω πως δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό και πρέπει αυτό το πρόβλημα να το έχουμε υπόψη μας. Ο Μάρκος Πίπερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και πολύ σύντομα. Αναφερθήκατε στις απαιτήσει που διατυπώνονται για τα νέα έργα, ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, οριμότητα και βιωσιμότητα. Αυτό ακριβώς περιγράφει και το Connecting Europe. Η διευκόλυνση συνδέωση στην Ευρώπη. Ρωτώ λοιπόν εάν στην πορεία αυτήν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις από το κράτη-μέλη για το πώς θα διαμορφωθούν οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί και πώς θα είναι συμβατοί με τα νέα μέτσα. Ευχαριστώ κύριος Μαρινέσκου. Thank you, President. Thank you, Commissioner. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για την ε, εισήγησή σας. Η ερώτησή, μας είναι, ερώτησή μου είναι θα έρθείτε ενώπιον του Κοινοβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού για το ΣΥΕΦ γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές αυτή τη στιγμή. Καταρχήν τα χρήματα αποφασίσαμε σε, σε σχέση με ένα ποσό, με, τώρα είναι διαφορετικό. Αποφασίσαμε σε σχέση με έναν κατάλογο σχεδίων και τον προορισμό τους, τόπο σιδηροδρόμους. Ενώ τώρα μας παρουσιάζεται ένα κατάλογο πρόγραμμα, ε, σχεδίων και μάλιστα να σας πω ότι εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε να παρουσιάσετε εσείς η Κομισιόν όλα τα προγράμματα που ζήτησαν τα κράτη-μέλη, γιατί χρειάζεται διαφάνεια. Εσείς λοιπόν αναφέρετε άλλα προγράμματα, τελείως διαφορετικά από αυτά που αποφασίσαμε τον κανονισμό. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, θα πρέπει να έρθετε ενώπιον του Κοινοβουλίου με την τροποποίηση του κανονισμού. Ευχαριστώ η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ανησυχία μου, διότι είχαμε 30 δις ξεκάθαρα και ξεκάθαρα όλα τα έργα και τα νούμερα ήταν ξεκάθαρα και τα έργα ήταν ξεκάθαρα. Τώρα με το σχέδιο Juncker ε, υπάρχουν διάφορα ρίσκα, διάφορα κίνδυνοι. Ε, ελπίζω αυτό να μην οδηγήσει σε τροποποιήσει τη συμφωνία μα, γιατί χρειάστηκε πολύ κόπος να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Αποκλείεται λοιπόν το δημόσιο χρέο. Για μα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάτε για όλη τη συγχρηματοδότηση ή μόνο για το 10%. Μπορείτε να το εξηγήσετε γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Είναι πολύ σημαντικό για την Ισπανία αυτό. Και επίση αύριο θα παρουσιάσετε στο Συμβούλιο ένα κατάλογο έργων. Η καταληκτική προθεσμία όμως είναι 26 Φεβρουαρίου του 2015. Ε, τι συμβαίνει, εσείς το έχετε κλείσει το θέμα, δίνουμε την ημερομηνία και εμψυχώνουμε τον κόσμο να παρουσιάσει έργα μέχρι την, 26, η Φεβρουαρίου και λέτε ότι δεν θα δώσετε τεχνική βοήθεια. Ποιο θα αξιολογήσει όμω και θα συμβουλεύσει για το κατά πόσο πραγματικά υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ο Ιβο Μπέλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κυρία Επίτροπε στο κέντρο. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Το έθεσαν οι διάφοροι συνάδελφοι. Συμφωνείτε μαζί μας, είναι προτεραιότητα για σας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι. Είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίζετε μαζί με τους συναδέλφους σας για τις κοινωνικές υποθέσεις, τους αρμοδίους επιτρόπους. Δεύτερον, το Port Package 3 έχει κολλήσει προς το παρόν. Περιμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ε, κρατικές ενισχύσεις από τον αρμόδιο Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό. Πώς θα προχωρήσετε ε, με αυτό το φάκελο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, Επίτροπε. Βρίσκομαι εδώ πίσω. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι δεν συμμεριζόμαστε από τον ενθουσιασμό σας ε, όσον αφορά το πρόγραμμα του Juncker, διότι δυστυχώς είναι προφανές ότι πρόκειται για μια επιχείρηση ε, ε, χρηματοδοτικής μηχανικής. Τα χρήματα αυτά είναι ανύπαρκτα και οι εγγυήσει που δίνονται δεν είναι πιστικές για μας. Είναι πολύ εύκολο να πολλαπλασιαστούν. Αν είναι τόσο εύκολο βάλω να πολλαπλασιαστούν έτσι εύκολα τα χρήματα, γιατί περιμέναμε πέντε χρόνια ενώ διάφορες χώρες βυθίζονται στην απελπισία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τούτου λεχθέντο. μπορείτε ίσω να το διαβάσετε στον Πρόεδρο Γιούνκερ. Τώρα όσον αφορά τι μεταφορέ, μιλήσατε για προτεραιότητα σε προγράμματα με καλή κοινωνικο-οικονομική απόδοση. Υπάρχουν όμω προγράμματα όπου επιμένετε, ε, ενώ ε, μελέτε έχουν αποδείξει ότι δεν θα έχουν κοινωνικο-οικονομική απόδοση. α πούμε το Ρήνο Λιών, ε, η ροή τη κίνηση διαρκώ μειώνεται, οπότε ελπίζουμε πω κάποια στιγμή θα λάβετε υπόψη αυτέ τι. Ε, μελέτες και θα το βάλετε στην άκρη. Ευχαριστώ. Ε, Μάτις Φον Μπιλτενμπούργκ. Ο Μάτις Φον Μπίλτεμπουργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη η πρόκληση για μας να συνεργαστούμε μαζί σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Όμως, ως προς τα νέα μέσα χρηματοδότησης επενδύσεων, Κάναμε συζήτηση για την αξιολόγηση εκ των προτέρων της ενδυνάμει αξιοποίησης των ε, χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο ε, της, ε, του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα μας οδηγήσει σε ανάπτυξη, ελπίζουμε. Ερωτώ όμως το εξής. Οι συγκεκριμένες ανάγκες του εκάθος του εκάστοτε έργου θα έχουν την πρωτοπορία όταν αξιοποιούμε τα διάφορα μέσα, ε, τα χρηματοοικονομικά και χρηματοδότησης. Πώς αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε και να το σιγουρέψουμε τελικά δεν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο χρηματοδότησης ή επένδυσης που να ε, κάνει τα έργα τόσο περίπλοκα ώστε ε, να ε, τελικά να προσκρούσουν πάνω σε τροχοπέδι. Ενδεχομένως αυτή είναι η περίπτωση του Άμστερνταμ και της αποβάθρας εκεί του υδατοφράκτη. Επόμενη βουλευτής. Ε, είμαι βουλευτής από την περιφέρεια του Λονδίνου και μπορώ να σας πω τι κάνουμε στο Λονδίνο για την ε, κινητικότητα μέσα στο άστι και για τις προσβάσιμε μεταφορές. Ωστόσο προτιμώ να μιλήσω για την οδική ασφάλεια. Ε, δεν νομίζω ότι με ικανοποιούν ιδιαίτερω αυτά που είπατε. Για παράδειγμα, έχουμε του πεζού. Το 1 το το θανάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι θάνατοι πεζών. Λέτε ότι δίνετε ε, προσοχή στους πολίτες. Πώς επιτρέπετε όμως ε, στα κράτη-μέλη να ξεφεύγουν με αυτό το μορατόριο για, τις μεγα... για τα μεγάλα οχήματα και ε, για τα HGV, τα τέτοιου είδους τεράστια φορτηγά, heavy good vehicle δηλαδή. Και έχουμε και θανάτους ποδηλατών. Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανονιστικές διατάξεις για αυτά τα τεράστια φορτηγά. Το κόμμα των εργατικών έχει δεσμευθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε και να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα λίγων ε, κατασκευαστών και λίγων ε, με που τους αρέσει να φωνασκούν χωρίς όμως να νοιάζονται για τους λαούς. Ευχαριστώ. Επόμενος βουλευτής, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο κυρία Μπούλτς και έχω δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Πρώτον, για το καμποτάζ. Εγώ είμαι από την Πολωνία και έχουμε 24% μερίδιο στο καμποτάζ σε όλη την Ευρώπη. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα του αθέμη του ανταγωνισμού και του κοινωνικού dumping. Είναι θέματα που έχουν θέσει οι κάτω χώρες, η Γαλλία και το Βέλγιο. Η Γαλλία ζητά αλλαγές στους κανονισμούς. Τι θα γίνει με την εναρμόνιση των ε, κανονισμών για τα εργασιακά, για τα κοινωνικά θέματα. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη να επέλθουν τέτοιου είδους αλλαγές. Και ποια είναι η γνώμη σας για τις πρόσφατες διατάξεις, τους κανονισμούς δηλαδή, σε σχέση με το χρόνο εργασίας και τον χρόνο ε, ε, ξεκούρασης ή αναψυχής των οδηγών φορτηγών. Είναι πράγματα που έχει υιοθετήσει πρόσφατα η Γαλλία και το Βέλγιο. Και τέλος για, την, για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ε, ε, ε, παίρνετε το χρόνο από τους άλλους. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Ελπίζω ότι στη διάρκεια των πέντε ετών της θητείας σας θα έχουμε καλή σχέση. Ναι, εδώ είμαι. Ε, στα, στα αριστερά σας. Η πρώτη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι αυτό που αναμένω από εσά, δεδομένου ότι είστε πολύ ισχυρή γυναίκα, προέρχεστε από το τομέα των επιχειρήσεων, είναι να δώσετε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις μεταφορές, στις υποδομές. Ο τομέας των μεταφορών δημιουργεί ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο και οι επενδύσεις αυτές στις μεταφορές θα πρέπει να είναι προτεραιότητα στο σχέδιο Juncker. Δεύτερον, όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη, ε, ε, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει περισσότερο να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι στη Ρουμανία όποτε θέλετε. Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια καλή διασύνδεση για τις περιφερειακές περιοχές. Ας πούμε, τις τουριστικές περιοχές που είναι υπέροχες ε, στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχουν μεταφορές, δεν υπάρχουν προσβάσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε, είμαι εδώ. Μιλήσατε κι εσείς ε, για το μέλλον της Λευκής Βίβλου, ότι δεν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε αναθεώρηση. Το είχατε πει παλιότερα αυτό, ισχύει ακόμη. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω για τους αερολιμένους που βρίσκονται σε ε, δυσκολίες ε, και προσπαθούν να εξασφαλίσουν μέσα από έναν ενιαίο ε, χώρο των εθέρων ή των αέριων μεταφορών επαρκή ε, κάλυψη. Μια τρίτη ερώτηση. Θα προσπαθήσετε να προχωρήσετε σε μια εναρμόνιση του ευρωπαϊκού συστήματος των διοδίων και δεν δεν αφορά μόνο τα γερμανικά διοδία. Σα ευχαριστώ. Εγώ επιμένω σε ένα ερώτημα που ήδη υπέβαλαν άλλοι συνάδελφοι. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια υποτίμηση του θέματο τη αστική κινητικότητα. Το 2050 το 82% του ευρωπαϊκού πληθυσμού θα ζει στις μετροπολιτικές περιοχές. Κινδυνεύουμε να φαινόμαστε σαν αριανοί. Μιλάμε για μεγάλα προγράμματα, μεγάλου άξονες, ενώ κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα που επικρατεί στι πόλει μα. Συζητάμε για το ETS, για την καταπολέμηση τη ρήπα, για τι κλιματικέ αλλαγές και δεν παρεμβαίνουμε εκεί όπου είναι απαραίτητο και επίγον να παρέμβουμε. Αυτή είναι, υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα μεγάλα διεθνή προγράμματα και τις παρεμβάσεις στις αστικές περιοχές που πρέπει να είναι προτεραιότητα και δεν θα γίνει προτεραιότητα αν το σχέδιο Juncker δεν προσγειωθεί να λύσει το πρόβλημα της ευελιξίας και το, της εθνικής χρηματοδότησης στα τοπικά προγράμματα και παρεμβάσεις. Ευχαριστώ. Can I ask if you've been involved in the UK's new road fund? Κυρία Σέμα, Μιλάτε για το σχέδιο υποδομών, όμως για τις παραβάσεις μήπως θα έπρεπε να εγκατασταθούν περισσότερες κάμερες. Ξέρετε όμως ότι είναι κατά της, η πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών και κυρίως των μεταφορέων. Δεύτερον, μιλάτε για χρήματα, αλλά βασικά μιλάτε για τα προγράμματα. Ε, πώς μπορείτε να δαπανάτε αυτά τα χρήματα πράγματα τόσο μάταια, ενώ ο προηγούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνε πολύ μεγάλα σφάλματα, ο προϋπολογισμός των μεταφορών. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Επίτροπε. Σίγουρα είναι εξαιρετική ιδέα το να συμμετέχει και να συμμετέχουμε στις επισκέψεις σας στις χώρες μας γιατί και από την πλευρά των υποδομών θα ήταν κάτι τέτοιο πολύ χρήσιμο. Όμως το κοινωνικό dumping δεν είναι κάτι που περιθωριακά συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξάλλου καθημερινά αυξάνεται ο αθέμητος ανταγωνισμός στον τομέα αυτό. Οι Υπουργοί των Μεταφορών οφείλουν πραγματικά να θέσουν τέλος στο κοινωνικό dumping και εσείς θα πρέπει να παίξετε ρόλο σα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Συγχαρητήρια για, και πολύ καλή επιτυχία ευχόμαστε για την σκληρή δουλειά που έχετε αναλάβει. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω εάν βλέπετε πρόβλημα στο να υπάρχουν διαφορετικές, ε, διαφορετικά στήματα προς την ασφάλιση των ε, ε, φορτηγών. Επίσης θέμα που αφορά την ασφάλεια στις μεταφορές και νομίζω ότι με αυτά κάλυψα το χρόνο μου. Κυρία Βοζενπέλη. Καλωσορίζω και εγώ κυρία Επίτροπε. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στα ποια θεωρείται σημαντικότερα έργα υποδομής στον Ανατολικό Διάδρομο, το Διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου που έχουν προστιθέμενη αξία για το κεντρικό δίκτυο. Και η δεύτερη, εάν σκέπτεστε μια προ, ε, εμπροστοβαρή χρηματοδότηση ή αντίθετα το, τη μείωση του κόστους της εθνικής χρηματοδότησης για τα έργα υποδομή, για την υλοποίηση των έργων υποδομή στι χώρε που βρίσκονται σε κρίση και ακολουθούν πρόγραμμα δημοσιονομική προσαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η σειρά μου τώρα τελευταίος. Και μετά εσείς θα έχετε το δύσκολο καθήκον να απαντήσετε. Λοιπόν, είπατε ότι δεν μπορείτε να τοποθετηθείτε για τα διόδια στη Γερμανία. Έστω. Αλλά καταρχήν, συμφωνείτε να υπάρχει μια βινιέτα η οποία επιβάλλει να πληρώνει το ίδιο και αυτός που χρησιμοποιεί πολύ το όχημά του και αυτός που το χρησιμοποιεί λίγο. Είναι οικολογικό, δεν είναι οικολογικό, είναι οικονομικό, δεν είναι οικονομικό κτλ. Για δε, συγγνώμη, την ε, Γερμανία, το να χρεώνει λιγότερο τον Γερμανό είναι διάκριση ή δεν είναι. Αυτό δεν είχε γίνει το 2009 ε, με τον ε, Τσίμερμαν Πρέπει να απαντήσετε τώρα, έστω και αν δεν ξέρετε τα συγκεκριμένα σχέδια, καταρχήν που στέκεστε. Και επίσης για τις θέσεις εργασίας, πώς μπορείτε, μάλλον για τα 100 εκατομμύρια που χρειάζονται από το Βερολίνο για την Πρατισλάβα. Πώς μπορείτε να υποχρεάσετε την, ε, στα επόμενα χρόνια τη Γερμανία να τα διαθέσει και να προχωρήσει στο έργο αυτό. Είναι θέσεις εργασίας αυτό. Το τούνελ στις Άλπεις. Το να μπει δηλαδή ένας, ε, ε, ένα τρυπάνι και να ανοίξει σύραγγα μέσα στις Άλπεις. Είναι θέση εργασίας. Τα 5-10 χιλιόμετρα που λείπουν έχουν προσθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Είναι αυτοπροτεραιότητα. Μια σειρά λοιπόν να ερωτήσει για σας και με χαρά και αδημονία περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Νομίζω ότι πρέπει να έρχομαι πιο συχνά να σας επισκέπτομαι στην Επιτροπή Μεταφορών, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις σας και πολύ λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμως και θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Μισό λεπτό παρακαλώ. 10 Δέκα λεπτά μου δίνουν. Ε, ελπίζω ότι δεν θα τα ξεπεράσω θα κάνω ό,τι μπορώ. Εν πάση περιπτώσει, θα απαντήσω γρήγορα σε όλη αυτή την πλειάδα ερωτήσεων που μου έχετε θέσει και ελπίζω να σα ικανοποιήσω αρκετά ώστε να με ξανακαλέσετε. Καταρχά για τα 300 δι, γιατί πάρα πολλοί ρωτήσατε για αυτά τα περιβόητα 300 δι. Να σα πω εξ αρχή ότι βεβαίω. Ε, ε, ε, σέβομαι τα χρήματα των φορολογουμένων. Εγώ ίδια έχω πληρώσει πάρα πολλούς φόρους και έτσι γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Αναφέρθηκα στα ιδιωτικά κονδύλια που κάθονται και περιμένουν μέχρι ότου να βγουν τα έργα για να μπορέσουν να επενδύσουν οι επενδυτές. Υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια επενδυτών που περιμένουν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να τα φέρουμε στο παιχνίδι. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτό το ταμείο με τα 300 δις. Από εκεί και πέρα, καλό είναι το ερώτημα σας. Όντως υπάρχει χρόνος για όλα τα πράγματα και όλα έρχονται όταν οριμάζει η στιγμή και ο χρόνος για να έρθουν. Μπορεί και άλλοι να είχαν σκεφτεί αυτό το ταμείο στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν τολμούσε να το προτείνει και να κάνει αυτό το βήμα. Τώρα έχουμε αυτό το τολμηρό βήμα με τη νέα πρόταση για τα 300 δις. Όντως είναι πολύ τολμηρό το βήμα, αλλά είναι απαραίτητο για να ε, σπρώξουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βρει καλύτερους μηχανισμούς και συνεχίζουμε να τους αναζητούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ανάπτυξη, αλλιώς η Ευρώπη θα γίνει μια ε, γριούλα η οποία θα κουνιέται στην πολυθρόνα της μόνο και θα περιμένει κάποιον να της φέρει το τσάι. Θα πρέπει λοιπόν κάτι άλλο να κάνουμε, κάπως αλλιώς να λειτουργήσουμε για να αναπτυχθούμε με παλμό, με, με, ζωντάνια, για να καινοτομήσουμε και να είμαστε εταίρος σημαντικό στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα. Αυτά καταρχάς, γενική δήλωση. Μπαίνω τώρα σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που μου έχουν τεθεί. Κύριε Φώστερ, μιλήσατε για την αεροπλοεία. Θα, σίγουρα θα το γνωρίζετε, ωστόσο Ποτέ δεν υπήρχε ε, στρατηγική βίβλος ε, για τα θέματα της αεροπλοείας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς θα το κάνουμε. Δεν λέω ότι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη χάρτα, αν θέλετε, που θα περιλαμβάνει τη στρατηγική μας για την αεροπλοεία μέσα σε ένα χρόνο, αλλά θα γίνει στη δική μας θητεία και σας καλώ να συμβάλλετε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στρατηγικές γραμμές, τη χάραξη της στρατηγικής καταρχάς για να ταυτοποιήσουμε τις ανάγκες και μετά να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις αεροπορικές εταιρείες, τις ευρωπαϊκές ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας είπα ότι ε, έχω συναντηθεί με όσο το δυνατόν περισσότερους και μεγαλύτερους εκπροσώπους ε, του κλάδου και με ενθαρρύνουν του κλάδου της αεροπλοείας όταν συζητώ μαζί τους αυτά τα θέματα και τους εξηγώ τις προθέσεις μας. Κύριε Βαντάλεν, μιλήσατε για τα εκοκόμπι, για αυτά τα πολύ μεγάλα ε, φορτηγά Ελπίζω να υπάρξει καλή συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και να γίνουν αυτά κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Ξέρω ότι ήταν αυτό πράγματι σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμη να διευκολύνει, να κάνει το παν για να υπάρξει συμφωνία. Εμείς επιθυμούμε τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, για το τέταρτο σιδηροδρομικό ε, πακέτο. Είμαι πεπισμένη και μάλιστα ελπίζω και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα σημειώσει πρόοδο σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες Έχουμε, δεν θα πρέπει όλο το πακέτο να μείνει πίσω. Ε, θα πρέπει το τεχνικό σκέλος να συνεχίσει να προοδεύει. Αλλά εμείς θέλουμε το πολιτικό να συμβαδίζει με το τεχνικό σκέλος. Γιατί υπογραμμίζω με όλους του, τους τόνους και με όλα τα χρώματα το πολιτικό να πηγαίνει δίπλα πλάι-πλάι με το τεχνικό. Υπάρχει τεχνολογία Και ο δεύτερος πυλώνας μας φέρνει τους επιχειρηματικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να εμπλέξουμε και να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία. Εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε και τα δύο σκέλη να συμβαδίσουν. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές. Αλλά ε, μέχρι τότε θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε όλα τα σκέλη του πακέτου της συμφωνίας να προχωρήσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτά μπορώ να πω για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ανησυχίες για ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταλαμβάνει τη θέση του οδηγού στην επιλογή των έργων. Και δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή ούτως ή άλλως. Θα συνεχίσω ε, σε μία άγουσα διαφανούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας με εσάς. Σε αυτό το σημείο όμως τονίζω για άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν θα βγει από αυτό το πακέτο. Απλά κάποια από τα έργα κάτω από την ομπρέλα του συνδέοντα στην Ευρώπη που μπορούν να χρηματοδοτηθούν με πιο φιλόδοξα ε, σχέδια επενδυτικά ή χρηματοδότησης, τότε θα γίνει αυτό και κάποια project πιο επικίνδυνα αν θέλετε, υψηλότερου ε, ρίσκου που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν βάσει του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη, τώρα θα μπορούν με τα νέα αυτά χρηματοδοτικά ή οικονομικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα τεθεί εν κινδύνο τίποτα από όλα αυτά που έχει υλοποιήσει ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη. Και το λέω ελπίζοντας ότι πραγματικά σας καθησυχάζω με τα λόγια μου αυτά. Και άλλωστε, ανοιχτός διαφανής διάλογος με εσάς. Αυτό θα έχω πάντοτε, δεν πρόκειται να κρύψω τίποτα. Και αν νομίζετε ότι κάτι σας έχει αποκριβεί, στείλτε μου ένα μήνυμα. Ε, έχω συνάδελφο που του έχω αναθέσει το καθήκον του συντονισμού των σχέσεών μας, ημώντε και ημών. Επομένως, θα δράσει ε, ε, κάθε φορά που θα μαθαίνει ότι οι ανάγκες σας δεν έχουν καλυφθεί. Θέλω να έχω έναν ανοιχτό, διαφανή, επικοδομητικό διάλογο μαζί σας. Πολλές ερωτήσεις μου τέθηκαν για το πακέτο των 3,3 δις. 3,3 δις από το συνδέονται στην Ευρώπη πήγαν σε αυτό το μηχανισμό επενδύσεων και χρηματοδότησης ε, για μόχλευση. Με μεγάλο ενθουσιασμό περιμένω όλα αυτά τα έργα. Γιατί έχουμε έργα που μπορούν να έχουν ένα λόγο ε, προσέλκυσης επενδύσεων 1 προς 5 ή 1 προς 15. Αλλά εάν τελικά δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο οποίο να θελήσουν να επενδύσουν οι επενδυτές, το να το δούμε αυτό, αυτό μιλάει από μόνο του. Εάν δηλαδή σε κάποιο project δεν βρεθούν καθόλου επενδυτές, τότε γιατί να θέλουμε εκεί να επενδύσουμε τα ε, χρήματα των φορολογουμένων. Ελπίζω ότι κάποια έργα πράγματι θα είναι ενδιαφέροντα και για την αγορά. Θα ε, καταφέρουν να ε, αναζωπυρώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και των επιχειρήσεων. Και όπως σας είπα, τα ταμεία συνοχής δεν τα αγγίζουμε καθόλου και πάρα πολλά έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτών. Τώρα, αποκλεισμό από το εθνικό έλλειμμα. Δεν είναι ε, αρμοδιότητά μου, όπως γνωρίζετε άμεσα. Τις επόμενες εβδομάδες θα εξηγηθεί λεπτομερώς το θέμα αυτό από τον κύριο Ντομπρόφσκι και θα υπάρξει επίσημη δήλωση από πλευρά του και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ιδαλλιώς ευχαρίστω ε, θα επανέλθω στην Επιτροπή σας και θα το εξηγήσω πώ ακριβώς θα γίνει μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες. Τώρα, κρατικές ενισχύσεις για τους λιμένες. Τι μπορώ να πω γι' αυτό. Χρειαζόμαστε τους κανόνες διαφάνειας που περιλαμβάνονται στις προτάσεις για τους λιμένες και αυτή τη μάχη θα δώσουμε. Θα μας βοηθήσει αυτό να ελέγχουμε καλύτερα τις κρατικές ενισχύσεις και θα ενθαρρύνουμε έτσι την ε, πιο ενάρετη κατανομή δημοσίων κονδυλίων. Θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι το κλειδί ε, που ε, δίνει απάντηση σε πάρα πολλές ερωτήσεις σημαντικές. Από εκεί και πέρα, ε, μου τέθηκε ερώτηση για την οδική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, ανά πάσα στιγμή, η οδική ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δεν κλείνει ποτέ. για όσο χρόνο κρατάει η θητεία μου στη θέση του Επιτρόπου για τις μεταφορές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Δεν μπορώ να σας πω ε, σε ποιο εξάμεινο θα γίνουν αυτά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ασχοληθούμε ιδιαίτερος με το θέμα. Δεν θα υπάρξει νέα λευκή βίβλος, ωστόσο θα κάνουμε τη σωστή αναθεώρηση των υφιστάμενων κειμένων, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις αλλαγές στις προτεραιότητες και ε, τις αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης του θέματος για να μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό παραδοτέο. Δεν θα είναι όμως αυτό το 2015. Όμως ένα από τα εξάμεινα της θητείας μας θα ε, αφιερωθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Και κύριε Κράμερ... Τώρα πρέπει να θυμηθώ τι με ρωτήσατε. Δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Mm, okay, I hope... Uh, λοιπόν, ελπίζω να κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Διορθώστε με παρακαλώ. Λοιπόν, ο Ριπένον πληρώνει και ε, ε διαχείριση αποβλήτων distant based charging, ε, χρέωση με βάση την απόσταση που διανύει κανείς και την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Αυτά μας ενδιαφέρουν κυρίως και έχουμε και το Eurovinet για τα οχήματα, τα αυτοκίνητα. Η εμπειρία που είχαμε με τα φορτηγά ήταν εξαιρετικά θετική και θέλουμε αυτό να το ε, επεκτείνουμε. Άλλωστε, το Eurovinet μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορες προκλήσεις. Δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Ωστόσο, ορισμένα κρατημέλη ε, και διάφορες ενώσεις και οργανώσεις μας ενθαρρύνουν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άκουσα την παρέμβασή σας απευθείας στα γερμανικά που μιλήσατε και αν τα κατάλαβα καλά... Ε, μπορείτε να το επαναλάβετε, θέλετε να κάνετε δήλωση για τη γερμανική προσέγγιση. Ναι, γιατί στη Γερμανία το 1992 η κυβέρνηση θέλησε να επιβάλλει διόδια στα φορτηγά περιορίζοντας τη φορολογία αντίστοιχα. Το απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, όπως και το 2004. Έτσι λοιπόν τώρα έχετε ε, αποφασίσει να το δεχθείτε αυτό ή θα κοιτάξετε να το αλλάξετε. Καλώς λέει η Επίτροπος. Ίσως να μην σας ικανοποιήσω ιδιαίτερως με την απάντησή μου, ωστόσο πραγματικά έχω την εντύπωση ότι οφείλω να υπερασπιστώ ε, με κάθε τρόπο τις βασικές αρχές των ευρωπαϊκών συνθήκων. Δεν είμαι νομικός και γνωρίζω ότι εάν κάποιος θέλει να αποφύγει κάτι, τότε μπορεί να βάλει ό,τι θέλει μέσα στις συμβάσεις και στις ρήτρε. Επομένως, θα διαβουλευθώ με τους αρμοδιούς και νομίζω ότι το κείμενο θα συνάδει με τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς το λύνει το ζήτημα ε, το κείμενο που θα προταθεί. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση έναντι αλλοδαπών σε σχέση με τους γηγενείς. Ε, ελπίζω και οι Γερμανοί να το λύσουν το θέμα αυτό, όμως εγώ καλούμε να προστατεύσω την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να επανέλθω και να απαντήσω σε κάποια άλλη στιγμή, όταν μάθω ακριβώς τι έχουν στο μυαλό τους, γιατί πολλές είναι οι εκδοχές που προβάλλονται, οι προτάσεις, αλλά δεν έχει έρθει τίποτα μπροστά μου ε, να το δω συγκεκριμένα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Είστε εδώ. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Και βεβαίως περιμένουμε να σας ξαναδούμε στο μέλλον. Θα σας προσκαλέσουμε και πάλι και σας ευχαριστώ για τη δέσμευση ότι θα ξανάρθετε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μπούλτς. Ήταν όντω μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Και θέλω να εισακούσετε αυτή μου την έκκληση. Θέλω να επενδύσουμε σε ενέργεια, γνώση, το χρόνο αυτό που έχουμε στη θέση μας να τον αφιερώσουμε σε προτάσεις που θα γίνονται και δεκτές. Ευχαριστώ. Να μην χάνουμε ενέργεια δηλαδή και χρόνο σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.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 So, Σας παρακαλώ πολύ όποιος είναι να μείνει μέσα να καθίσει στη θέση του ή δάλλως να φύγει από την αίθουσα. Να ξεκινήσουμε παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση εφαρμογής για την εισαγωγή εφιών συστημάτων μεταφορών. Δίνω το λόγο στην ε, κυρία Κοψίνσκα από την Επιτροπή. Ε, το λόγο. Ήσασταν και χθες εδώ, μας γνωρίζετε πια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα σας. Ναι, ήμουν εδώ και το πρωί και άκουσα τη συζήτησή σας με την Επίτροπο Μπούλτς. Ίσως ε, δεν ετέθησαν πολλά ερωτήματα για το ITS επειδή μου τα φυλάγατε εμένα. Ε, πολύ ευχαριστώ λοιπόν να σας απαντήσω όταν έρθει η ώρα. ITS, FEE, συστήματα μεταφορών. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το πακέτο και την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας ITS και του προγράμματος δράσης το 2008 το Δεκέμβριο ξεκίνησε υιοθετούμενη η οδηγία μαζί με 24 δράσεις Στοχευμένε έξι τομείς προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας της οδηγίας. Αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την νομοθετική διαδικασία, με την τροποποίηση της οδηγίας, αλλά αυτό ήδη προβλεπόταν εξ αρχής και στόχος είναι η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της των διεπαφών, της διεπαφικότητας της ε, μεταφοράς. Ήθελα να πω ότι είχαμε μια πολύ κατακαιρματισμένη εξέλιξη στο τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ένα μέρο τη Ευρώπη θεωρεί ότι είναι πολύ καλέ εξελίξει και γρήγορε, ενώ άλλο μέρο θεωρεί ότι βράδυ μπορούμε σε σχέση με την ανάπτυξη των εφιών συστημάτων μεταφορών και την εφαρμογή του. Το Αύγουστο του 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή με ένα καλό ε, παράδειγμα της εφαρμογής ε, και της συνεργασίας των συνομοθετών, το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, εξασφάλισαν την ταχεία και πρόσκοπτη εφαρμογή, έγκριση, συγγνώμη, και την πρόοδο στον τομέα των ευφυών συστημάτων. Οι στόχοι της οδηγίας είναι η επιτάχυνση της συντονισμένης ανάπτυξης και χρήσης των ευφυών συστημάτων στους δρόμους, αλλά και το, η διασύνδεση με τους λοιπούς τρόπους των μεταφορών. Η συνέχεια λοιπόν και η διεπαφή επαφή σε όλη την Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αυτής της ε, και ήταν η πρώτη, αν δεν το πολύ πολύ δεύτερη οδηγία η οποία αξιοποίησε ένα νέο μέσο των κατεξουσιοδοτησεων πράξεων, οδηγία η οποία επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει με τις, να βελτιώσει με τις κατεξουδότητες συμπράξεων την ανάπτυξη των ε, ITS. Επτά έτη λοιπόν έχει διάρκεια η εντολή αυτή, πάει μέχρι το 2017 και η έκθεση την οποία έχω έρθει να σας παρουσιάσω αφορά μια δέσμη ε, προτάσεων προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την υλοποίηση της οδηγίας ITS και των κατεξουδότησης πράξεων, αλλά και έγγραφο εργασίας του προσωπικού για την πρόοδο της χρήσης του προγράμματος ε, δράσεως για το ITS, αλλά και ένα άλλο έγγραφο συμπληρωματικό, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί ενημέρωση για την πρόοδο, με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών, όπως ήταν υποχρεωμένα να καταθέσουν δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δηλώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης για το ITS και να περάσω μετά στην έκθεση σε σχέση με την περιγραφή του προγράμματος δράσεως. Είναι αρκετά πλήρης περιγραφή των ε, όσων έχουν εξασφαλιστεί στο χώρο του ITS με 24 δράσεις, τους 6 τομείς προτεραιότητας. Επίσης, εξετάζεται η βελτίωση της ε, συνειδητοποίησης και αναγνώρισης του συστήματος ευφυών μεταφορών, πώς γίνεται το κύριο σύστημα μεταφορών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επισημαίνονται ορισμένα ζητήματα που παραμένουν και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. Η αναγκαιότητα, παραδείγματι, για, την, ε, για το ρήμα της πρόσβασης στους πολιτουργικούς τρόπους μεταφορών, και μεταφορά δεδομένων, η ανάγκη για εργασία σε ένα στονισμένο τρόπο, στους πολιτουργικούς τρόπους μεταφορά και επίσης την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ε, κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο ώστε να καλύπτουμε και το μηχανισμό αλλά και τον ορίζοντα 2020 ανάλογα με τη χρήση των ε, κονδυλίων για το ITS. Σε σχέση με την έκθεση τώρα για την οδηγία, στόχος της ήταν η ανάλυση του πώς λειτουργεί η οδηγία, πώς η πρόοδος έχει επιτευχθεί και τι ακόμα μένει να γίνει. Και θα είμαι ειλικρινής. Ήταν περίπλοκο το μέσον ακόμα και όταν ε, προτείναμε εμείς την οδηγία, γνωρίζαμε ότι ε, πιάναμε ένα τομέα πολύ ευαίσθητο τεχνολογικά με πολλές αλλαγές και ριζικές αλλαγές, ταχύες αλλαγές και γι' αυτό θεωρούσαμε ότι η κατεξουσιοδότηση πράξη θα είναι η καλύτερη για να μην πω η μόνη δυνατότητα που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε τις ε, τόσο ταχείες μεταβόλες στον τομέα αυτών. Θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους μέσα και μηχανισμούς μπορούμε να έχουμε ένα καλό εργαλείο Μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τους ειδικού από τα κράτη-μέλη αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα στην ομάδα εργασία για τα OFES, σύστημα μεταφορών, γιατί υπενθυμίζω ότι η οδηγία ITS δεν δίνει εντολή για ανάπτυξη του συστήματος εφιών μεταφορών, αλλά λέει ότι μέσω των κατεξουσιοδότησης πράξεων μπορούν να υπάρξουν, μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και διατύπωση απαιτήσεων, άπαξ και αναπτυχθεί σύστημα ευφυών μεταφορών, η ευφυές σύστημα μεταφορών. Ε, αυτό στον τρόπο με τον οποίο μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, γιατί κράτη, κάποια κράτη-μέλη στα οποία ήδη υπήρχαν ε, μηχανισμοί ευφυών μεταφορών. Τώρα, και από τις συζητήσεις με τους ιδιώτες φορείς. Και από τις γενικότερες επαφές μας βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό προϋποθέσεων και προδιαγραφών στους τομείς όπως έχουν αυτές συμφωνηθεί και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και προς τις ε, προδιαγραφές και προς τη λειτουργικότητα με συγκεκριμένες επιλογές εφόσον συμφωνήσουμε πού θέλουμε να πάμε και αυτό μπορεί να γίνει συνεργατικά και όχι να κάθεται η Επιτροπή σε μια γωνία για να ορίζει προδιαγραφές για το ITS. Επίσης θεωρούμε ότι μπορεί να επιτρεπεί μια πολύ αναλογική προσέγγιση, άρα να μην γίνει υποχρεωτική ανάπτυξη του συστήματος επιμεταφορών, αλλά ε, να προχωρήσουμε με συμφωνίες άπαξ και υπάρξουν σχετικές εξελίξεις. Οι δράσεις προτεραιότητας όπως αυτές περιγράφονται στην οδηγία ε, χαίρουν τώρα ενός πλήρου συνόλου οργανωτικών διατυπώσεων που υποστηρίζει και ο τομέας των μεταφορών και τα κρατημέλη και βέβαια γενικός στόχος καινοτομία και ψηφιοποίηση μεταφορές προδιαγραφές έχουμε για τα, τους διάφορους τομείς, για την ασφάλεια ε, και για την πληροφορία σχετικά με την οδική ασφάλεια που παρέχεται στους χρήστες δωρεάν. Τέλος, έχουμε ε, προβλέψεις για το, ε, για το και για, συγκεκριμένα για το οίκο, για το Ευρωκοινοβούλιο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόθεση αυτής της υπηρεσίας ε, επίγουσες ανάγκες στο ηλεκτρονικό τηλέφωνο ε, ή call ώστε να αναβαθμιστεί το θέμα της ασφάλειας και σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνεται και στην πρόταση για μεταρρύθμιση της, ε, του κανονισμού περί έγκρισης τύπου Α. Και να ευχαριστήσω την κυρία Σενάλοβα για την εργασία της επ' αυτού και σας συγχαίρω για τα αποτελέσματα που επιτύχατε. Τέλος, πληροφορίες πραγματικής ε, ε, ε, μάλλον κυκλοφορίες σε πραγματικό χρόνο. Εδώ σας ενημέρωσα ήδη τον Οκτώβριο κατά εξοδότηση πράξη που προβλέπει για τις προδιαγραφές για την παροχή πληροφοριών κυκλοφορίας, κυκλοφοριακής κίνησης μάλλον σε πραγματικό χρόνο. Ελπίζω πως θα έχετε την επίσημη έγκριση, την επίσημη μάλλον υποβολή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Ένα σχόλιο για ένα θέμα που δεν αντιμετωπίσαμε και αυτό είναι η συγκεκριμένη χώρη στάθμευσης, ασφαλούς στάθμευσης για τα φορτηγά. Στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας το είχαμε συζητήσει, ωστόσο ε, το συζητήσαμε και με τα κρατημέλη και με τον ε, εκπροσώπους του κλάδου και επίσης δώσαμε πληροφορίες σχετικά στην Επιτροπή Μεταφορών και αποφασίσαμε ότι για την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου τομέα. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να το θέσουμε σε αναμονή. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε εάν αλλάξουν τα δεδομένα από πλευρά κρατών μελών και από πλευρά του κλάδου, ότι υπάρχει δυνατότητα και ότι υπάρχει σχετική σχετικός χώρος στην αγορά για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος κράτηση χώρου στάθμευσης. Ε, τώρα, να σας πω για ποιον θεμάτων δεν δουλεύουμε. Καταρχήν, ε, ε, υπηρεσίες ενημέρωσης για τις πολυτροπικές μεταφορές είναι το τελευταίο και πιο δύσκολο κομμάτι γιατί αφορά μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων καθώς και φορέων που εμπλέκονται. Ξεκινήσαμε την εργασία μας γιατί χαρακτηριστικά αυτό το μήνα. Πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους των κρατών μελών έγινε τη παρουσία ενός συναδέλφου από την ε, γραμματεία της Επιτροπής Μεταφορών, όπου αρχίσαμε να συζητούμε τους ορισμούς καθώς και τις ανάγκες των χρηστών. Αυτό που θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε μέσω των χαρακτηριστικών είναι τα στοιχεία πολυτροπικών μεταφορών, για την κυκλοφορία και για τη μετακίνηση με ελαφρύς ε, τρόπους όπως ας πούμε ποδηλασία, συγκεκριμένη σταθμή ή νέες υπηρεσίες ε, ε, κινητικότητας όπως τα κοινά αυτοκίνητα, τα το car sharing, μοιρασιά δηλαδή ενός αυτοκινήτου. Αυτά λοιπόν μέσω της οδηγίας ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στο πιο δυναμικό εργαλείο της κατεξουδότησης πράξης ώστε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου νέες τεχνολογικές λύσεις αλλά όχι μόνο τεχνολογικές λύσεις, νέες, ε, νέα σχήματα κινητικότητας, νέες μορφές κινητικότητας δημιουργούνται ή εν πάση περιπτώσει αναζωογονούνται κάθε χρόνο. Ελπίζουμε ότι με, αυτές τις με αυτήν την κατεξοδότηση πράκτηνη η ολοκλήρωση των, μεταφορών, των, των υπηρεσιών μεταφορών και καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δυνατοτήτων με όλους τους τρόπους μεταφορών θα διευκολυνθεί. Επιπλέον, διότι δεν ήταν ένας από τους τομείς προτεραιότητας, ε, της δράσης προτεραιότητας στην οδηγία, αλλά ήταν ε, ε, μία από τις δράσεις στο πρόγραμμα δράσης και για αυτήν είχαμε μεγάλη ενθάρρυνση καθώς και ε, αιτήματα από το κλάδο και από τα κράτη-μέλη για τα συστήματα συνεργασίας, ιδιαίτερα η επικοινωνία ανάμεσα στα οχήματα και τις υποδομές. Διότι αυτό είναι κάτι που πριν από έξι χρόνια, όταν ξεκινήσαμε την οδηγία και το πρόγραμμα δράσης, εξακολουθούσε να είναι στον τομέα του απόμακρου μέλλοντος. Αυτό σήμαινε μεγάλη συμμετοχή των, ε, των ε, ενδιαφερομένων από το κλάδο και θέλαμε να φτιάξουμε ένα οδικό χάρτη, μια στρατηγική για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη στο πλαίσιο της ανάπτυξης του CITS. Ήδη γνωρίζουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα υπό εξέλιξη τα περισσότερα κράτη-μέλη εξετάζουν τι πρέπει να γίνει ώστε να καταστεί πιο ευφυής ε, η υποδομή τους ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό η επικοινωνία ανάμεσα στα οχήματα και τις υποδομές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί η χωρητικότητα των δικτύων. Και έπειτα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα των συνδεδεμένων οχημάτων όσο και σας φαίνεται αυτό παράδοξο, ώστε να εξισορροπηθεί εκ νέου η χρήση των διαφόρων τρόπων. Πολύ συχνά ο κόσμος μένει στο αυτοκίνητό του γιατί δεν ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει τρόπο μεταφορών, ότι μπορεί να αφήσει το μάξι του κάπου ας πούμε, και να συνεχίσει με διαφορετικό τρόπο ε, να συνδεθεί ολόκληρο το σύστημα μεταφορών λοιπόν όσον αφορά την χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών για τους χρήστες και τους ε, οδηγούς και τους επιβάτες. Τώρα, θα δείτε επίσης μια αξιολόγηση των χρηματοδοτικών πόρων που χρειάζονται και που ε, ε, χρησιμοποιούνται. Εδώ έχουμε σχετικά πρόσφατα χαρακτηριστικά και δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού αντίκτυπου μιας ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα. Αλλά ελπίζουμε όπως είπα στην αρχή, ότι στον σχεδιασμό τα ευφύ e, αυτά συστήματα μεταφορών είναι στον, ε, στους στόχους και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα αναπτύξουν ιδέες σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί. Στην έκθεση, και αυτή θα είναι η τελευταία μου δήλωση, στην έκθεση επίσης εξετάσαμε τους, ε, τα όρια της οδηγίας και καθώς και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι το ITS, αν και αρχικά αφορούσε μόνο το οδικές μεταφορές ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και κάποια οριζόντια θέματα, σίγουρα αυτά που σχετίζονται με την πρόσβαση και την διαθεσιμότητα για τη μεταφορά δεδομένων. Ή, ανέκαθεν λέγαμε ότι το θέμα της προστασίας των δεδομένων θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και έχει γίνει αυτό για όλα τα χαρακτηριστικά. Επίσης τώρα ξέρουμε και βλέπουμε τι, να, τι μπορεί να γίνει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα συστήματα σχεδιασμού και επίσης εφόσον ε, εκπνέει το χρονικό διάστημα ε, της ε, ανάθεσης κατά εξουσιοδότηση το 2017 θα κάνουμε μια εκτίμηση για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και εάν ε, ισχύει κάτι τέτοιο, το 2016 θα υποβάλουμε νέα πρόταση. Πάντως τώρα θα ξεκινήσουμε τον μελέτη αντικτύπου και θα ήταν πρόημο τώρα να ε, προβλέψουμε οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντερκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Θεωρώ όμως ότι έχουμε ώρα ε, ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτό κάνουμε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως λέει ο Πρόεδρος. Καλώς. Τότε θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ευχαριστώ βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ σαφή της παρουσίαση. Εμείς στη πολιτική ομάδα του ΕΛΚ Πράγματι θέλουμε έξυπνα, καθαρά και ανατόμα συστήματα μεταφορών. Θεωρούμε ότι αυτό βοηθάει την Ευρώπη να κινηθεί προς τα εμπρός. Και καλώς υπάρχει το ITS, το έξυπνο σύστημα μεταφορών. Όμως είναι ένα project το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη ορατότητα. Ίσως διαβάζω λάθος ιστοσελίδες και λάθος δημοσιεύματα. Μπορείτε να πείτε δύο λόγια για την ορατότητα αυτού του έργου και ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Και δεύτερο ερώτημα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ινδία και στην Κίνα. Από το σημείο εκκίνησης ξεκίνησαν γρηγορότερα όσον αφορά σε αυτόν τον αγώνα για τα νέα έργα, δημιουργώντας συνδέσεις, ε, κόμβους το καθεξής. Νομίζω ότι η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά αργή. Και από εκεί και πέρα, ο Γαλιλαίος, το σύστημα Γαλιλαίος, τι κάνουν τα αρμόδια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτό. Ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και για το πασίγνωστο Google. Την περασμένη εβδομάδα υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για το Google. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχει εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορισμένα σχόλια να κάνει για το έξυπνο σύστημα μεταφορών και την Google. Και στη συνέχεια για τα διόδια στην Ευρώπη. Είδαμε την Επιτροπή Μεταφορών στις κατοχώρες την περασμένη εβδομάδα και συνεχίσαμε να βλέπουμε ε, φορτηγά με πέντε ε, σήματα ε, ευρωπαϊκά, πέντε αστέρων σήματα κυκλοφορίας. Ειδικά σε θέματα αστικής ευθύνης, ευθύνης γενικότερα και ασφάλισης. Τι μπορείτε να μας πείτε. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αργεί και αυτό καθυστερεί ε, την ε, έλευση της τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σέρτογκ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Πολύ διαφωτιστικά. Και έβηχα. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης. Διαπίστωσα ότι οι επιχειρήσεις κράτησης και εξασφάλισης ασφαλών και προστατευμένων θέσεων εργασίας για φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα δεν χρήζει περαιτέρω χειρισμών. Έτσι λέτε. Για μένα αυτό είναι το μέσο ο παρουσιάζει μεγαλύτερες ανάγκες. Διότι ιδιαίτερα σε χώρες ε, διέλευσης οι περιοχές διέλευσης, οι χώροι στάθμευσης έχουν πια φτάσει στο αδιαχώρητο. Στην ε, Γερμανία οι ε, οδηγοί αναγκάζονται να παρκάρουν στην ε, λωρίδα έκτακτης ανάγκης πάνω στο δρόμο γιατί δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις στους χώρους στάθμευσης. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει ιδιαίτερα να παρακολουθήσουμε και τις περαιτέρω, ε, να παρακολουθήσουμε το τομέα αυτών, γιατί είναι κέρια σημασία για την παραπέρα εξέλιξη και ανάπτυξη ενός συστήματος ευφυών μεταφορών. Γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση. Ευχαριστώ. Αυτά είδαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ. Στα αγγλικά. Λέτε ότι θα θέλατε να επιταχύνετε τη διαδικασία της εφαρμογής του συστήματος ε, των, ε, του συστήματος μεταφορών Βλέπουμε ότι σε ορισμένους τομείς υπάρχουν εξελίξεις ταχύτερες, ενώ αλλού είναι βραδύτερες, σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, πού συγκεκριμένα θέλετε τη δική μας υποστήριξη. Επίσης μιλήσατε για τα κατεξουσιοδότηση συμπράξης για να επιτέχει τη διαδικασία. Πότε θα έχουμε τις πρώτες κατεξουσιοδότηση συμπράξης επί τάπητος, για να δούμε ακριβώς τι ζητάτε. Και τρίτον, πολύ απλά, επίσης, πολύ σημαντικό όμως για εμάς τους φιλελευθέρους, ε, για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τι κάνετε, διαρκώς ενημερώνεστε, ενημερώνετε δηλαδή τις προτάσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Έχω ένα στρατογικό ερώτημα να θέσω για το θέμα αυτό. Με την παρουσίασή σας είδαμε ότι θα αναπτυχθεί το FES σύστημα ε, μεταφορών και αυτό και από πλευράς υποδομών και από πλευράς υπηρεσιών θα είναι ε, καθοριστικό στοιχείο για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Όμως, ε, συζητώντας με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς και με άλλους αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατάλαβα ότι ε, μένει μεγάλη απόσταση να διανύσουμε. Δεν έχουν μπει ακόμα τα θεμελιώδη για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Το, αυτό το σχέδιο θα το ε, ε, ενσωματώσετε στην ενία ψηφιακή αγορά. Θα έχετε ε, τις απαραίτητες κανονιστικές διατάξεις αλλά και τα απαραίτητα χρήματα. Π.χ. στο μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένοι φάκελοι αναθέμα, μεταφορές, ψηφιακές πλατφόρμες και ενέργεια, για παράδειγμα. Και πράγματι έχετε δίκιο, έχουμε οριζόντιες προτεραιότητες σε όλα αυτά και στο μηχανισμό γιατί συνδέοντας την Ευρώπη όταν ε, ικανοποιούνται δύο διαφορετικά κεφάλαια ε, προτεραιοτήτων, δικαιούται κανείς μια περαιτέρω επιδότηση, αν θέλετε, μια περαιτέρω ενίσχυση, ένα μπόνους. Άρα, αυτά που λέτε μπαίνουν οριζόντια, θα άπτονται περισσότερο ε, ανώτερων του ενός ε, ε, κεφαλαίων και άρα θα υπάρξει πόνους. Και με τη δεδομένη τη σημασία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ε, και από τη στιγμή που θα έχουμε και επενδύσεις και υπηρεσίες, ποιος θα είναι ο καθοδηγητής αν θέλετε όλων αυτών. Οι μεταφορές πώς θα ωφεληθούν επειδή θα ενσωματωθούν στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Το ερώτημα ε, για τη Google είναι ψηφιακής φύσης. Σε κάθε περίπτωση οι μεταφορές ε, μιλούν για το STI, για το Intelligent Transport System, είναι όμως και αυτόνομες. Δεν, δεν μιλήσατε καθόλου για αυτά, ούτε ε, και η Επίτροπος μίλησε για αυτά. Δηλαδή, νομικά και τεχνικά πώς θα αλληλοσυνδέονται και θα διαρθρώνονται αυτά τα θέματα. Οι μεταφορές είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό από το ψηφιακό κόσμο και πώς θα ενσωματωθεί στις γενικές πολιτικές για την ψηφιακή εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάμε τον κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την έκθεση, για την οδηγία που μπαίνει τώρα έτσι στο, στην πολιτική αντιπαράθεση. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας μίλησε με τρόπο πολύ γενικό και τυπικό σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι πολύ περιορισμένη η συμβατότητα. Έχουμε να κάνουμε με ένα ε, ε, μοσαϊκό ή με μία κουρελού η οποία έχει πολύ διαφορετικά κομμάτια μη συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ε, μιλάμε επί παραδείγματι για την Ευρωβινιέντα όπως σήμερα και μιλούμε για τέλος ανάλογα με την χρήση που θα επιβάλλεται για την χρήση των του οδικού δικτύου. Μιλούμε για συμβατότητα στο τέταρτο πακέτο σιδηροδρομικό, ε, των σιδηροδρόμων, για την ένταση του ρεύματος ή για την χρήση σημάτων φωτεινών ε, και άλλων συστημάτων που θέλουμε να ενσωματώσουμε που είναι τόσο διαφορετικά από, την, το ένα κράτος στο άλλο. Και βλέπουμε ένα άλλο σύστημα, το σύστημα των εφιών μεταφορών. Ένα ακόμη διαφορετικό σύστημα με πάλι διαφορετική εικόνα κράτος μέλος. Άκουσα κάποιες παρατηρήσεις για τα συστήματα των διοδίων μέσα στην Ευρώπη ε, που μας παρουσίασαν οι εμπορογνώμονες όταν είχαν έρθει από την ε, θέση του ομιλητή να μας ε, εξηγήσουν πόσο μόνο το δικό του σύστημα, το ιταλικό ήταν, το γερμανικό ήταν, το γαλλικό ήταν, είναι το ευφιέστερο και το πιο πρακτικό και το πιο καλό αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη. Και σε αυτό πρέπει να συζητήσουμε ουσιαστικά και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά όπως και με τις ε, προτάσεις που μας παρουσιάστηκαν τώρα. Γιατί έχουμε 8 δις ευρώ επενδύσεις στο Γαλιλαίος επί παραδείγματι. Ντομινίκ από τη Γαλλική Γουιάν, Γουιάννα, από υπερπόντια γαλλική κτήση εστάλει δορυφόρος στο διάστημα. Πολύ ωραία. Κάλυψη. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα, ξέρουμε τι θα κάνει, θα καταγράφει προσωπικά δεδομένα του κάθε ενός εξημών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων και τους εκπροσώπους των κρατών μελών να κάτσει και να αποφασίσει και ενδεχομένω να ιδρύσει μία ομάδα η οποία θα έχει και μεγάλους παραγωγούς όπως Alstrom, Siemens, Bombardier και ποιου άλλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών γιατί έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας με την Airbus. Με την Airbus δεν θα, χωρίς την Airbus δεν θα είχαμε ποτέ ε, μπορέσει να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό των Αμερικανών εάν δεν ήταν μια λογική και καλή συνεργασία βιομηχανιών της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και εδώ ακριβώς έχουμε να κάνουμε με αυτές τις έννοιες που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξισώσουμε, δηλαδή να καταστήσουμε συμβατά τα συστήματα το μεν με το δε. Μιλούμε για κλιματικές αλλαγές, ο καθένας Γράφεται στον κατάλογο των ομιλητών, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να το αποφύγω, αλλά θα αναγκαστώ να το πω τελικά, γιατί τελικά αυτό που κάνουμε είναι μια κατακριματισμένη δράση. Λίμα, Φερρυπίν, πάμε ε, ε, να πούμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τι εκπομπέ οξυδίου του άνθρακα, αλλά τι πιο πολλέ εκπομπέ οξυδίου του άνθρακα τι έχουμε από τι ε, συμφορήσει τι κυκλοφοριακέ ε, και από άλλα ζητήματα στα οποία δεν έχουμε μπορέσει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αυτό πρέπει να καταστήσουμε μεταξύ μα συμβατό και σε αυτό ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε και από την Επίτροπο Μπόλτς ε, πιο συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Έτσι μόνο μπορούμε να είμαστε και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί. Ευχαριστώ που με αφήσατε να ξεπεράσω το χρόνο μου. Αλλά όφιλα να το πράξω. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Με χαρά σας ακούσαμε και πάλι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και διαθυξικεδαστικό. Ναι, μα είναι τόσα πολλά που ε, βρίσκονται σε διαρκή κίνηση κτλ. Παρακαλώ, η επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαιρετική της παρουσίαση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω μοιάζει με αυτό του συναδέλφου Κάμπη, ο οποίος πήρε το λόγο προλίγου. Δηλαδή, σε θέματα έξυπνου συστήματος μεταφορών, όντως η Ευρώπη είναι ουραγός, καθυστερή. Κι όμως, Έχουμε πάρα πολλές γνώσεις, έχουμε εξαιρετικές υποδομές, έχουμε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις ε, πηγαίνουν αλλού σε άλλα μέρη του κόσμου για να δοκιμάσουν τις ε, καινοτόμες τους ιδέες στην Καλιφόρνια, των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Κίνα, αλλού. Σε κάθε περίπτωση δεν δοκιμάζουν τις ε, ιδέες τους στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να νομοθετεί πιο έξυπνα. Έχουμε το Smart Regulation και καλώς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια που πρέπει επιτέλους να καταρριφθούν έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να καινοτομήσουν στην Ευρώπη και να ε, ε, δοκιμάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους εδώ στην Ευρώπη. Γνωρίζετε ποιες είναι οι διατάξεις που ε, παρεμποδίζουν τις επιχειρήσεις και δεν τους επιτρέπουν να ε, καινοτομήσουν εδώ, από εκεί και πέρα. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από πλευρά ε, έξυπνου συστήματο μεταφορών συγκριτικά με την Κίνα και τι ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζετερκόχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω και εγώ μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ενδιαφέρει ο συσχετισμός μεταξύ εφιών συστημάτων μεταφορών και ηλεκτρονικού συστήματος συνδυασμού μεταφορών. Έχετε κάποια δουλειά ήδη ξεκινήσει το με αυτόν ή τίποτα ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Σλάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση και την ε, επίκληση του ονόματός μου. Θα ήθελα να φερθώ προς το θέμα της ε, εισαγωγής του e-call. Έχει κρατήσει τρία χρόνια, ήταν εντατική η δουλειά. Έχουμε κάνει έκθεση ιδέας πρωτοβουλία στην Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών και με συνεισηγητή τον κύριο Κόχ ο οποίος ασχολείται με διάφορα συγκεκριμένα θέματα και την προετοιμασία των υποδομών και το καθεξής. Αυτή η δραστηριότητα, επιβεβαιώνω και εγώ, ήταν αρκετά περίπλοκη και παραμένει. Η συνεργασία λοιπόν της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εσωτερικής Αγοράς ε, ε, και πολιτικών ελευθεριών ήταν πολύ σημαντική και εδώ θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί όταν έρθει η ώρα να εγκριθεί το σύστημα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και τη προστασία του, στον βαθμό που αυτά καλύπτονται, στο σύστημα e-call ηλεκτρονικής πλήσης. Εμείς υποστηρίξαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σύστημα αυτό και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και στην κοινή γνώμη πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί. Η ερώτησή μου λοιπόν έχει να κάνει και με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Πρέπει και αυτή να την προετοιμάσουμε και να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία ώστε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεργασία τους Ευχαριστώ πολύ. Άλλος ένας στον κατάλογο των ομιλητών και είναι ο υποφαινόμενος με τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς ε, για το σύστημα στάθμευσης για τα ε, φορτηγά. Όταν είχε ξεκινήσει η ιστορία για, τους, για τα φορτηγά στη Γερμανία, ε, ήμασταν κατά διότι λέγανε η Γερμανία ότι ήταν ελληματικό το σύστημα των των χώρων στάθμευση για τα φορτηγά κατά 14-15 θέσεις στη Γερμανία και όταν ήρθε η ιστορία με τα gigaliners, με τα πολύ μεγάλα φορτηγά, το επιχείρημα ήταν ότι αυτά πιάνουν και δύο θέσεις φορτηγών, οπότε είναι ακόμα πιο μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα λοιπόν μας λέτε ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται, δεν χρειάζεται να μελετήσετε περαιτέρω το ζήτημα και ενώ βλέπουμε ότι θα οξυνθεί περαιτέρω με τα γίγα το πρόβλημα της στάθμισης των φορτηγών, μας λέτε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επίσης, σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Κούν, έχει βγει τώρα, αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της συνεργασίας χάρη στην, Air, στην οποία προχώρησε η Airbus, μπορούμε να δούμε αντίστοιχα και το TGV και το ICE και το ελβετικό τρένο και το Ιταλικό. Το καθένα για διαφορετικά χαρίσματα. Ε, οι Ελβετοί έχουν ακρίβεια, οι Ιταλοί έχουν κομψότητα, οι Γερμανοί έχουν αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, είναι δυνατόν κάθε σύστημα να είναι διαφορετικό. Φυσικά η βιομηχανία έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την ποικιλία. Το είδαμε άλλωστε. Όταν κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε μία ε, μηχανή η οποία να μπορεί να σύρει διαφορετικά τρένα ανάλογα με τη χώρα. Ούτε μία για 10.000, για 10 χιλιόμετρα δεν μπορούσαμε να βρούμε μία μηχανή που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Προφανώς και τη βιομηχανία τη συμφέρει αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε το σύστημα της ε, ακύρωσης εισιτήριων όταν είναι κανείς στο εξωτερικό ξέρει πολύ καλά ότι τελικά δεν θα χρησιμοποιήσει εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς γιατί αλλού πρέπει να το χτυπήσει το εισιτήριο πριν να, βγει, πριν μπεις ε, στο τραμ, αλλού πρέπει να αγοράσει το εισιτήριο μέσα, ε, αλλού πρέπει να το έχει αγοράσει από το περίπτερο και το καθεξής. Ξέρουμε ότι στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά αυτών που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο. Λοιπόν, 10 λεπτά γιατί έχω καλή διάθεση λόγω και Κιάκη Βασίλειου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Είναι αδύνατο να απαντήσω μέσα σε 10 λεπτά, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εκτιμώ ιδιαίτερο το μεγάλο πλήθος των ερωτήσεών σας, γιατί δείχνει πόσο σας συναρπάζει αυτό το πεδίο. Κάτι το οποίο συναρπάζει βεβαίως και εμάς. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις, μήπως κερδίσω έτσι κάπως περισσότερο χρόνο. Να ξεκινήσω από την ερώτηση του κυρίου Βαντερκάμπ. Την ορατότητα του εφιού συστήματος μεταφορών. Νομίζουμε ότι το έχουμε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι όταν μιλούμε για ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και υποδομές θα πρέπει το ευφυές σύστημα μεταφορών να αποτελεί μέρος τους και έχουμε ειδικό άρθρο στον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα μεταφορών, τον κλάδο των μεταφορων τέν TEN-T. Πρέπει να είναι σαφές ότι εξετάζουμε τις επενδύσεις στις υποδομές. Δεν πάμε σε μη έξυπνες υποδομές και μετά να προσθέσουμε το έξυπνο σκέλος, γιατί αυτό δεν μας βοηθάει. Αναπτύσσοντας το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη και το ten ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το σκέλος των μεταφορών, θα δείτε ότι ε, το FES σύστημα μεταφορών θα γίνεται όλο και πιο πολύ streamlined, θα μπαίνει όλο και πιο πολύ ε, στο επίκεντρο, αν θέλετε, όλων των δράσεων. Και έχουμε διάφορα φυλάδια και δημοσιεύσεις και δημοσιεύματα, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό. Ε, τέθηκαν ερωτήματα για τα ηλεκτρονικά διόδια, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας του Γαλιλαίου ε, σε σχέση με το σύστημα εφιών μεταφορών. Θα θυμάστε ότι τα ηλεκτρονικά διόδια στην Ευρώπη διέπονται από διαφορετικά νομοθετήματα από τη στιγμή που έχουμε και απόφαση και οδηγία. Και υπ' αυτή την έννοια ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει με το θα θέλαμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, εμείς θα επιθυμούσαμε ένα ενιαίο και μοναδικό σύστημα ηλεκτρονικό και να εισπράττονται τα διόδια παντού στην Ευρώπη μέσω αυτού του συστήματος και έτσι τα φορτηγά καταρχάς και αργότερα η, τα γιοταχή ε, ε, ε, να μπορούν να μην να μην χρειάζεται, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουν διάφορα και περιπλόκα συστήματα. Ωστόσο, Υπάρχουν διάφορες ομάδες εμπλεκόμενων φορέων και αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο να γίνει προς το παρόν. Πού μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο, με ρωτήσατε. Θέλουμε να μας στηρίξετε για να προωθήσουμε αυτή την έννοια, την αντίληψη της αξιοποίησης της τεχνολογίας για να οδηγήσουμε και να μετακινηθούμε καλύτερα σε όλη την Ευρώπη. Μιλούμε επίση για την ασφαλή και σίγουρη στάθμευση. Μου θέσατε τέτοιου είδου ερωτήματα και εσεί, Πρόεδρε, μεταξύ των άλλων συναδέλφων σα, να σα υπενθυμίσω ότι στην οδηγία έχουμε περιλάβει την ασφαλή, την επαρκή στάθμευση, ε, την διαθεσιμότητα των πληροφοριών για αυτούς τους χώρους στάθμευσης και τη δυνατότητα κλεισίματος θέσης. Και υπάρχει κατεξουσιοδότηση ε, πράξης σχετικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρεί τα κρατη με μία ενιαία ευρωπαϊκή πύλη, σημείο εισόδου αν θέλετε, με πληροφορίες για τους χώρους στάθμευσης. Ε, μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα χωρητικότητας βεβαίως και δυναμικού, έτσι. Αυτό το συνειδητοποιούμε. Ωστόσο, ένα σύστημα που θα λειτουργεί σωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα κάνει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης να, να αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Γιατί αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι υπάρχουν καινοί χώροι στάθμευσης σε ένα μέρος και υπερσυγκέντρωση ε, οχημάτων σε άλλο μέρος για να σταθμεύσουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η σωστή διευθέτηση, χωροταξική αν θέλετε διαρρύθμιση των χώρων στάθμευσης για τα φορτηγά. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι έχουμε τρεις ε, ε εξουσιοδοτήσει πράξεις έτοιμες, σχεδόν τέσσερις θα έλεγα και η πέμπτη ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Ε, άλλο ερώτημα μας ε, τέθηκε. για τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται η γενοποίηση των μεταφορών με το ΕΦΙΕ e σύστημα μεταφορών στην ευρύτερη ημερήσια διάταξη για την ψηφιακή εποχή, την ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Να σας πω ότι σε όλες τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέκαθεν το θέμα αυτό είναι παρόν. Συζητούμε, όπως είπε και η Επίτροπος, το πρόγραμμα εργασιών, το οριστικοποιούμε για την επόμενη χρονιά, το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα σας το παρουσιάσουμε λίγα συντόμω και μέρος του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η υποβολή νομοθετικής ε, ε, πρότασης για πρόσβαση σε δεδομένα ε, που έχουν να κάνουν με τα ταξίδια και τις μεταφορές. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος μεγάλη σε σχέση με την Ευρώπη από τη μία και τα άλλα μέρη του κόσμου από την άλλη. Ορισμένοι είπατε ότι ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λειτουργεί ως τροχοπέδι στη διαδικασία. Αυτό είναι το σχόλιο σας. Εγώ δυσκολεύομαι να απαντήσω από αυτού και να το σχολιάσω. Ε, καταλαβαίνετε. Ωστόσο, όταν βλέπουμε τόσο ευαίσθητα πεδία από πλευράς τεχνολογίας όπως είναι το σύστημα έξυπνων μεταφορών, τότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας και άλλα ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά, όπως είναι η προστασία των δεδομένων. Πρέπει να διαβουλευτούμε με τον ελεγκτή, τον Ευρωπαίο ελεγκτή αρμόδιο για τα ε, προσωπικά δεδομένα. Έχουμε ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, και μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει και μια συγκεκριμένη ομάδα ασχολείται με τα θέματα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ευθύνη ε, και πολύ σημαντικό θα είναι το θέμα της ευθύνης της διασυνοριακής. Εξετάζουμε τα διάφορα συστήματα συνεργασίας και γι' αυτό αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε πρώτα νομοθετική πρόταση, πρώτα να συγκεντρώσουμε τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς, τους εμπλεκόμενους φορείς, να συζητήσουμε με όλους αυτούς τους για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα σημαντικά ε, σημεία ε, πράγματι λαμβάνονται υπόψη και μετά να υποβάλουμε πρόταση νομοθετική για τα συνεργατικά συστήματα, τα συστήματα συνεργασίας. Και αν δείτε τις προτάσεις ε, του Αντιπροέδρου Άνσιπ και του Επιτρόπου Έτιγκερ σε θέματα ψηφιακά, θα δείτε ότι όλα αυτά ε, αφορούν και το θέμα των μεταφορών και του εφιού συστήματος μεταφορών, π.χ. διασυνοριακή πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αυτό, και εδώ απαντώ εν μέρη στο ερώτημα του Προέδρου, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν μιλούμε για πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, ταξιδιωτικές, π.χ. διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων, πληροφόρηση για τις υφιστάμενες διαθέσιμες τιμές ε, για τα εισιτηρία και το καθεξής ε, πληροφόρηση και πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις ταξιδιωτικές επιλογές. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της νομοθετικής πρότασης που συντάσσουμε αυτή τη στιγμή, που διατυπώνουμε. Και τέλος, εξίσου σημαντικό, πρόσβαση στην πληροφόρηση και στα στοιχεία. Τι θέλω να πω. Ε, παρουσιάσατε το παράδειγμα του Λονδίνου όταν συζητούσατε με την Επίτροπο προλίγου. Στο Λονδίνο αποφάσισαν να ανοίξουν όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τη μετάβαση. Δηλαδή όλα τα στοιχεία, όλες οι πληροφορίες για τις δημόσιες μεταφορές στο Λονδίνο είναι τώρα όλα αυτά διαθέσιμα, ανοιχτά. Και άρα έχουν αναπτυχθεί νέες υπηρεσίες πληροφόρησης, έχουν αναπτυχθεί από διαφόρους νέα εργαλεία που θα διευκολύνουν τον κόσμο να ε, κάνει την επιλογή του κάθε μέρα για τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθεί μέσα στην πόλη. Εμείς δεν κάνουμε όλα τα δεδομένα διαθέσιμα σε, στον οποιονδήποτε με εντελώς ανοιχτό τρόπο για άλλους λόγους. Και γνωρίζουμε ότι ορισμένες από τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και το, τα ταξίδια, τη μετάβαση στην Ευρώπη, οφείλονται στο γεγονός ότι ορισμένοι κλάδοι δεν είναι έτοιμοι να μοιραστούν στοιχεία και πληροφορίες για την εκάστοτε μεταφορά. Και με τη νέα νομοθετική πρόταση αυτό το κενό θα έρθουμε να καλύψουμε. Φιλοδοξούμε. Και ε, ένα σχόλιο να κάνω για το e-call, την ηλεκτρονική ε, κλήση. Ε, είναι περίπλοκη η πρόταση αυτή Πράγματι και δεν έχει έρθει στο κατάλληλο χρόνο. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε όλα αυτά. Θα είναι όμως ένα πρώτο παράδειγμα ενός συνεργατικού σχήματος μεταξύ κρατών μελών, γιατί βασίζεται σε στοιχεία που θα εκπέμπει το όχημα και θα συνδυάζονται αυτά τα στοιχεία με τα στοιχεία των υποδομών και των υπηρεσιών έτσι ώστε να υπάρξει άμεση βοήθεια σε περίπτωση επίγουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσίαση και για τις ερωτήσεις. Τελειώνει έτσι αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Έχουμε μια μικρή δεξίωση για τα Χριστούγεννα εδώ έξω. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Τα απόγευμα βέβαια. Ξαναρχίζουμε στις 3 με την ακρόαση για την σύνδεση στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.